Καθίστε παρακαλώ. Εγώ θα μιλήσω. Εδώ πριν από λίγο τελειώσαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ΑΦΚΟ, συνταγματικών υποθέσεων. Αλλά η Προεδρία είναι διπλή, γιατί είναι διπλή συνεδρίαση. Επομένως, θα δίνουμε το λόγο σε όποιον ε, ζητάει το λόγο, αλλά μία θα παίρνει ένας ε, από την Οικονομική Επιτροπή το λόγο και μία ε, θα την παίρνει από την ε, Συνταγματική Επιτροπή. Κάνουμε αυτή τη μεικτή συνεδρίαση λοιπόν και τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε σήμερα, τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι κυρίως οικονομικά θέματα, επομένως η βασική επιτροπή ας πούμε είναι η οικονομική. Αλλά πάντα τα οικονομικά προβλήματα συνδέονται με θεσμικά προβλήματα, επομένως και η Συνταγματική Επιτροπή εμπλέκεται. Επομένως η Συνταγματική Επιτροπή θέλει να παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή όσο μπορεί πιο επιμελώς τις ε, εργασίες για αυτή τη νέα συνθήκη. Τα θεσμικά προβλήματα συνδέονται με το γεγονός ότι πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη, διακυβερνητική συνθήκη και επομένως είναι θέμα που ενδιαφέρει την ε, Επιτροπή ΑΦΚΟ. Σήμερα νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε τους τρεις εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συνθήκη. Τον κύριο Μπροκ, τον κύριο Γουαλτιέρη και τον κύριο Φερχόφστακ. Ε, θα μας πούν τι επαφές είχαν μέχρι στιγμής και θα ακούσουμε κάποιους ε, προβληματισμούς των μελών της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Συνταγματικής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν ε, θα δούμε τι θα κάνουμε εφ' εξής. Κυρία Μπόλς, θέλει να πει και αυτή κάποια έτσι, εισαγωγικά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ στο χαρτί μου λέει ότι υπάρχει σχέδιο ημερήσιας διάταξης και λέω να την εγκρίνουμε αν κανείς έχει αντίρρηση. Σε αυτά που είπε ο κύριος Χασίνη έχω να πω μόνο ότι η, Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Νομισματική ασχολήθηκε με το εξάμετρο και μετά με άλλα δύο μέτρα, το δίμετρο και όλα πέρασαν πολύ ανώδυνα. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή τη νέα συνθήκη και είμαι σίγουρος ότι ο καθένας θα πει το λοκάκι του όπως πρέπει. Ας μην ξοδέψω άλλο χρόνο. Έχουμε όμως έναν κατάλογο ομιλητών με 19 ήδη ονόματα και οι υπόλοιποι θα εγγραφούν με οφθαλμοθυρία, catch Αλλά παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι και περιεκτικοί. Αυτή που είναι από την ΑΦΚΟ να κουνάνε το χέρι τους προς τη γραμματεία της ΑΦΚΟ και αυτοί που είναι από την εικόνα να κουνάνε το χέρι τους από την άλλη μεριά που είναι η γραμματεία της εικόνα. Έχουμε ήδη τους συντονιστές, για τους υπόλοιπους λέω, οι συντονιστές να μην κουνάνε. Λοιπόν, μήπως να αρχίσουμε με τον κύριο Πρόγκ. Ναι, νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Να ακούσουμε καταρχήν τους τρεις εισηγητές που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο. βλέπω τον κύριο Μπροκ, πρώτο και καλύτερο, και συνεχεί οι άλλοι δύο. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που έχουμε τόσο βραχυπρόθεσμα τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε αυτή τη συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Ε, Σήμερα έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασία και αυτό είναι καλό να ακούσουμε τις απόψεις σας και όχι να μας ακούσετε εσείς εμάς, για να ξέρουμε πώς εκτιμάτε την κατάσταση και πώς θα καταλήξουμε σε κάποιες διατυπώσεις που θα ικανοποιήσουν τους πάντες. Στη σημερινή συνεδρίαση, κατά βάση, έγινε μία δημοσκόπηση των αντιπροσωπιών, καταρχήν στις νέες χώρες που δεν είναι χώρες του ευρώ, που βρίσκεται η διαδικασία εκεί, ποιες είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά μέχρι στιγμή ε, όλοι είναι ευθυγραμμισμένοι και θέλουν να παραμείνουν ε, μαζί μας. Ε, η Μεγάλη Βρετανία μάλιστα ευχαρίστησε πολύ φιλικά για τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις συζητήσεις. Παρόλο βέβαια που τη ουσία δεν έχει συμβάλει σε τίποτα. Συνάδελφο Γκολτιέρη Φερόφσατ και ο υποφαινόμενο, έχουμε καθορίσει κάποια κεντρικά σημεία για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και τις ιδέες μας. Και θα ήθελα από αυτού να πω ότι βέβαια είπαμε όσον αφορά τους βασικούς στόχους Golden Pool δηλαδή και την αντίστροφη πλειοψηφία συμφωνούμε. αναρωτιόμαστε κατά πόσον αυτό θα πρέπει να περάσει σε αυτή τη συνθήκη και αν ναι υπό ποια μορφή. Παραδείγματο χάρη ρώτησα κατά πόσον αυτό που οι κρατών κυβερνήσεων ότι δηλαδή αυτή η συνθήκη θα πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να περάσει στην ε, συνθήκη της Ένωσης κατά πόσο θα μπορέσει αυτό να βγει από τις ιδεολογικές σκέψεις και να περάσει στα δεσμευτικά άρθρα της συνθήκης. Αυτές ήταν οι συστηματικές σκέψεις που ακούστηκαν, αλλά επί της ουσίας δεν είχε κανένας ουσιαστικές αντιρρήσεις. Οπότε θα ήταν δυνατόν να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, γιατί εάν με πρώτη ευκαιρία αυτό θα περάσει στη συνθήκη δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για συνταγματικά θέματα που θα επιδεινώσουν και θα καθαστήσουν πιο δύσκολη την μετάβαση αυτή. Και ε, θα πρέπει να προσέξουμε για να μην έχουμε προβλήματα με τη συνθήκη για το ευρώ και αυτή τη συνθήκη εδώ. Δεύτερο σημείο που παρουσιάστηκε σήμερα. Στο σχέδιο της συνθήκης αναφέρεται ότι εν τελευταία αναλύση το κοινοτικό δίκαιο θα υπερισχύει του διεθνούς αυτού δικαίου και ότι δεν θα επιτρέπεται να υποσκαπτεί όσον αφορά την ερμηνεία που θα δώσουμε. Εμείς θέλουμε να καθορίσουμε και μας υποστήριξαν πολλές αντιπροσωπείες πάνω σε αυτό ότι θα πρέπει να εγγραφεί ρητά ότι η δευτερογενής ε, νομοθεσία καταρχήν θα περάσει στην ε, κοινοτική νομοθεσία. Αυτό είναι ο κύριος κανόνας, ότι πρόκειται δηλαδή για κοινοτική απόφαση. Απ' την άλλη αυτό σημαίνει ότι δεν υποσκάλεται το δικαίωμα στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, όσον αφορά το λεγόμενο six-pack, καταστήσαμε απόλυτα σαφές ότι δεν επιτρέπεται να αποδυναμωθεί αυτή η νομοθεσία και επιβεβαιώθηκε αυτό και από τις νομικέ υπηρεσίες ότι μια τέτοια συνθήκη δεν δίνει τι νομικές δυνατότητε να, μην, να υστερήσουμε σχετικά με τη λύση του six-pack. Γιατί άμα διαβάσει κανένα το σχέδιο συνθήκη, θα δει ότι ορισμένε από τι απαιτήσει που αναφέρονται εκεί βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του six-pack ή κάτω από αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο, παραδείγματος χάρη όσον αφορά την αντίστροφη πλειοψηφία. Ή και όσον αφορά τις εξωτερικούς ελέγχους που πρότεινε η Κομισιόν τον Οκτώβριο. στον αφορα την ότι και αυτό είναι ένα επιχείρημα ούτως ώστε αυτά να παραμείνουν μόνο μέσα στα πλαίσια της κοινωτικής νομοθεσίας. Και θεωρώ, και νομίζω αυτό διαφαίνεται κιόλα, ότι αν πάρει κανένα συνθήκη, η συνθήκη αυτή δεν είναι εξίσου ισχυρή για να επιτευχθεί ο κοινοτικό στόχο. Αυτό είναι ένα θέμα που θίξαν πολλές άλλες αντιπροσωπείες. Εκπληκτικά μεγάλος αριθμός κρατών συμφωνούσαν μαζί μας πάνω σε αυτό. Οπότε και εδώ θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε να υπάρχει ένας πιο έντονος ορισμός εδώ. Και είναι καλό να δούμε ότι ακριβώς αυτές οι χώρες που θέλησαν ε, να αντιδράσουν στο Κοινοβούλιο όταν μιλούσαμε για την αντίστροφη πλειοψηφία στο Six park. Τώρα θέλουν να περάσει αυτό στη συνθήκη. Αυτή η χώρα που ξέρω καλύτερα αναφέρεται σε θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, ισορροπία μεταξύ των, ε, ε των χρεών κλπ. Και που τη διέγραψαν το 2005 τη διατύπωση αυτή από τη συνθήκη σταθερότητας, τώρα θέλουν να επανέλθει θα πρέπει να δούμε ότι και στο θέμα αυτό θα συζητήσουμε περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εμεί θέλουμε στα σημεία αυτά να ενδυναμώσουμε τη δευτερογενή ε, νομοθεσία και το six μπορεί να ενδυναμωθεί και ότι δεν πρέπει ποτέ να ειστερήσουμε σχετικά με αυτά που έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα γιατί αυτό θα το κατανοούσαν γλίγορα οι αγορές και αν καταλάβαιναν οι αγορές ότι αυτή η συνθήκη δεν οδηγεί σε περισσότερο έλεγχο αλλά σε λιγότερο, τι νόημα θα είχε. Γιατί θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και το θέμα αυτό του ευρωπαϊκά Δικαστηρίου που είναι πολύ πιο αποτελεσματικό για κάποια θέματα. Ο Ρομπέρτο θα το αναπτύξει αυτό. Και ένα άλλο σημείο όσον αφορά η ενδυναμωμένη συνεργασία. Και αυτό αναφέρεται στο άρθρο 10 της συνθήκης. Και είπαμε ότι εντάξει, αν υπάρχει θα πρέπει να το αναφέρουμε στα πλαίσια του άρθρου 20 της συνθήκης. Γιατί ακριβώς αυτό αναφέρεται και στην δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Και εδώ νομίζω μπορούμε επίσης να προχωρήσουμε. Letztlich Fragen stecken, die mit der Rolle des Europäischen Parlaments zu tun Αυτά έχουν όλα σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και το άρθρο 12 που ασχολείται με τα κοινοβούλια, με τις βουλές γενικά, όσον αφορά αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υπάρχει κάποια έκθεση, αντιαπλή ενημέρωση προβλέπεται και μια νέα συνένευση των ε, επιτροπών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών για οικονομικά ε, θέματα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό είναι προβληματικό, γιατί εδώ υπάρχουν διακανονισμοί που αφορούν το κοινοτικό ε, δίκαιο και οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου διακανονίζουν συνθήκη και θα πρέπει να βρούμε μια λύση παρόλη την αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν βέβαια τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό γίνεται μόνο μέσω του κοινοτικού δικαίου. Υπήρχαν και κάποιες ιδέες, πρέπει να συζητηθούν ακόμα πώς θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά θα πρέπει να είναι και σαφές ποιες είναι οι αρμοδιότητες πιανού βάζω τις συνθήκες, για να μην καταπατάτε κανένα δίκαιο. Σε γενικές γραμμές, θεωρώ ότι ένα μεγάλο αριθμό των αντιπροσωπιών υποδέχθηκε πολύ φιλικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέχρι στιγμή είχαμε ε, πολύ καλέ δυνατότητε και χάρη του ε, επικεφαλή των συζητήσεων να συμμετάσχουμε. Μέχρι τι 29 Δεκεμβρίου θα, 29 Δεκεμβρίου θα πρέπει να βάλουμε γραπτέ προτάσεις οι οποίε θα εξεταστούν στις 6 Ιανουαρίου σε μια δεύτερη συνεδρίαση με στόχο η ομάδα εργασίας να ολοκληρώσει εργασίες μέχρι τις 20 Ιανουαρίου πριν προωθηθεί το θέμα στο πολιτικό επίπεδο. Και γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα εισαγωγικά. Ε, όλοι θέλουμε να ακούσουμε σήμερα γιατί αύριο θα προσπαθήσουμε να κάτσουμε να καταγράψουμε κάτι για να είναι πιο σαφή τα πράγματα. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον απόψε ή αύριο το πρωί να έχουμε γραπτά τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων. Τι πιστεύουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε για να πληρώσουμε τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Ας ακούσουμε όπως είπα τους τρεις προσώπους και μετά τους υπόλοιπους. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί είμαστε εδώ κυρίως για να ακούσουμε τις συνεισφορές των μελών των δύο επιτροπών. Προσπαθήσαμε να σεβαστούμε τη βασική εντολή που μας έδωσε η διάσκεψη των Προέδρων, η οποία ήταν να εξασφαλίσουμε το σεβασμό της ε, κυριαρχίας του πρωτογενούς και δευτερογενούς ε, κοινοτικού δικαίου και να ενισχύσουμε και να μην ε, αποδυναμώσουμε το ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτή την εντολή προσπαθήσαμε καταρχήν να ζητήσουμε διευκρινήσεις για τους, τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Συνόδου ό,τι αφορά το πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο και τι μπορεί να εφαρμοστεί μέσω αυτού. Θέσαμε την ερώτηση αλλά δεν λάβαμε απάντηση. Ε, γιατί μας είπαν ότι η συνθήκη θα έχει συμβολικό χαρακτήρα ε, εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα θα μπορούσαν να είχαν γίνει, αν όχι όλα, μέσω τη δευτερογενού νομοθεσία. Επίση, εκφράσαμε ανησυχίε για τον κίνδυνο επικαλύψεων με τον, τους κανόνες και τις αρμοδιότητες ε, που προβλέπει το σχέδιο συνθήκης. Να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το άρθρο 3, που είναι η καρδιά αυτής της συνθήκης. Το άρθρο που μιλάει για το χρυσό κανόνα και τους μηχανισμούς που θα αρχίσουν να ισχύουν στην εθνική νομοθεσία. Διαφορετικά κατόφλια θα έχουμε από αυτά που προβλέπει το πακέτο των, των έξι νομοθετημάτων. Εδώ έχουμε ένα κατόφλι 0,5. Τελείως διαφορετικό. Το θέμα δεν είναι θέμα αριθμών, είναι και θέμα ποιοτικό. Γιατί το σύστημα που προκύπτει από αυτό το σχέδιο κειμένου στο άρθρο 3 είναι ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης. Δηλαδή, κάθε κρατός μέλος αξιολογεί μόνο του το δικό του κατόφλι και προσδιορίζει το κατόφλι και τις ε, συνθήκες υπό τις οποίες δεν το σέβεται. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση με αυτό που ισχύει σήμερα ε, για το ευρωπαϊκό σύστημα ε, παρακολούθησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Θέσαμε λοιπόν αυτό το θέμα παρότι δεν μπήκαμε σε συγκεκριμένη εξέταση του άρθρου 3, γιατί αφού το έγινε μια γενική συζήτηση, α, περάσαμε μόνο στην εξέταση του άρθρου 1 και εκεί σταματήσαμε. Εκεί θέσαμε κάποια ερωτήματα για το σύστημα εφαρμογής α, ε, τους, του σχεδίου συνθήκης, το οποίο είναι αδύναμο, γιατί βασίζεται μόνο ε, σε ένα άρθρο για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο είναι το άρθρο 273 της Συνδικής της Λισαβόνας, που είναι ένας ειδικός τρόπος χρήσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εγείρει νομικά προβλήματα. Ε, γιατί λέει το κείμενο ότι θα πρέπει να αναφέρεται σε θέματα που προβλέπει η συνθήκη, κάτι που δεν ε, ισχύει. Ε, και ότι θα εφαρμόζεται μέσω κυρώσεων. Έπειτα, ε, μιλήσαμε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είπε και ο κύριος Μπροκ, και όταν πέρασαμε στην ε, συγκεκριμένη εξέταση των άρθρων, είπαμε στο πρώτο άρθρο να υπάρξει μια αναφορά στην ανάπτυξη. Μια πρόταση που ε, υποστηρίχθηκε από όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες. Αλλά τελικά δεν έγινε δεκτή. Τη βάλαν σε αγγίλες. Θα περιμένουμε τον επόμενο γύρο συζητήσεων. Η εντύπωσή μου είναι ότι η όλη προσπάθεια θα μας πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε. Από ό,τι περίμεναν διοργανωτές τουλάχιστον. Τέλος, ο Ουίδων Φερχόστατ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως έχουν πει και άλλοι, εδώ ήρθαμε για να εξετάσουμε μαζί τη συμφωνία και να κάνουμε μια κοινή ανάλυση, να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ως προς το πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Όταν αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις το απόγευμα, είχαμε ρωτήσει γιατί χρειάζεται αυτή η συμφωνία. Εφόσον τα περισσότερα πόσα προβλέπει θα μπορούσαν να γίνουν με δευτερογενή νομοθεσία ή με βάση το άρθρο 136 της συνθήκης ή με την ενισχυμένη συνεργασία βάσει των άρθρων 326 με 334. Και μας απάντησε η νομική υπηρεσία το απόγευμα επαναλαμβάνω ότι σχεδόν τα πάντα θα μπορούσαν να γίνουν με δευτερογενή νομοθεσία σχεδόν, αλλά σχεδόν δεν θα πει όλα. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι σαφής απάντηση. Όλα μπορούν να γίνουν ή με ενισχυμένη συνεργασία ή με δευτερογενή νομοθεσία ή με το πρωτόκολλο 12 με συνδυασμό των τριών μεθόδων και με ρόλο και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Φαίνεται ότι είναι για πολιτικούς συμβολικούς λόγους που θέλουν να κάνουν τη συμφωνία έτσι. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος. Αν αρχίσουμε έτσι, τότε κάθε φορά θα υπάρχει ο πειρασμός να προστίθενται κεφάλαια Τώρα το λέμε για δημοσιονομική πειθαρχία και για τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 126, αλλά άμα γίνει αυτό και εγκριθεί θα αρχίσουν ξανά. Κάθε φορά που θα θέλουν να αναπτύξουν ή να εφαρμόσουν μια καινούργια πολιτική στο φορολογικό τομέα ή στον οικονομικό τομέα θα χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ο κίνδυνος του προηγούμενου δηλαδή. Πρέπει επομένως να κάνουμε μια επιλογή στρατηγικής σήμερα και τις επόμενες μέρες. Θέλουμε στενή συμφωνία που να περιορίζεται στα δύο συγκεκριμένα θέματα που αναφέρει το 126 προβλέπει συμφωνία μεταξύ χωρών μελών για να ψηφίσουν ομοιόμορφα όταν και τα λοιπά. Και μετά υπάρχει αυτό που προβλέπει το άρθρο 3. Θέλουμε λοιπόν ευρύτερη συμφωνία ή στενή. Νομίζω ότι εξαρτάται από το αν θα έχουμε την εγγύηση της βιωσιμότητας αυτής της συμφωνίας θα είναι αιώνια κτήμα ΕΣΑΗ e για τις επόμενες γενιές και τις επόμενες συμφωνίες ή μήπως θα προσθεθεί κάποιο άρθρο τελικά όπου αυτόματα όλη η συμφωνία θα μπαίνει, θα ενσωματώνεται στις συνθήκες αφού την εγκρίνουν βέβαια όλες οι χώρες μέλη ή μήπως μπορούμε να βάλουμε μια ρήτρα ηλιοβασιλέματος που λέμε. Μήπως θα ισχύει μόνο για ορισμένο αριθμό ετών και μετά πρέπει να επανέλθουμε να δούμε τι θα την κάνουμε. Αν θα μείνει έξω από τις συνθήκες ή αν θα μπει μέσα. Το πρώτο ερώτημα πρέπει εδώ να λύσουμε αν μπορούμε να βάλουμε ένα άρθρο όπου να διασφαλίζεται ότι σε κάποιο χρόνο όλα αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες συνθήκες και στο πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο, τότε ίσως πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία. Αν όμως δεν γίνεται να δοθεί αυτή η διαβεβαίωση ή εγγύηση, τότε νομίζω πρέπει να επιλέξουμε τη στενή έννοια της συμφωνίας αυτής. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Και το δευτέρο είναι ότι χρησιμοποιούν το 273 για να επιταχύνουν τη διαδικασία το οποίο δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί τα 60 χρόνια που υπάρχει η ΕΟΚ και η Ένωση. Μια φορά προσπάθησα ως Πρωθυπουργό να το χρησιμοποιήσω το 273 γιατί υπάρχει και μια διαφορετική ερμηνεία των οδηγιών γιατί τότε πρέπει να χρησιμοποιεί το 273 δηλαδή για θέμα που σχετίζεται μεν με τις συνθήκες αλλά υπάρχει κάποια διαφορετική ερμηνεία και τότε μπορεί σαν συμβιβασμό να το θέσει κανείς στα δικαστήρια. Είναι μάλλον άρθρο που χρησιμοποιείται μόνο για περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας που δίνουν ορισμένες χώρες μέλη. Μπορεί να αφορά οδηγία, μπορεί να αφορά οτιδήποτε άλλο. Όχι όμως για αυτό που το θέλουν τώρα. Τα άλλα άρθρα, 259 ας πούμε, χώρα κατά χώρας, διότι κάποια χώρα παραβιάζει τη συνθήκη, αυτό έχει χρησιμοποιηθεί έξι φορές σε 60 χρόνια. Και μετά υπάρχει βέβαια φυσικά και το 258. Όταν η Κομισιόν προσφεύγει κατά μια χώρα γιατί παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 2.000 φορές. Βλέπετε τη διαφορά λοιπόν. Κάτι που χρησιμοποιήθηκε 2.000 φορές και παραπάνω και κάτι που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται Βέβαια πολύ σπάνια και μια χώρα προσφεύγει κατά άλλη χώρα για παραβίαση τη συνθήκη ή του κοινοτικού δικαίου. Να, αυτά είναι τα ερωτηματικά που μας θέτει η χρήση του, 273. Γιατί κανονικά δεν αφορά καθόλου την Κομισιόν. Πώς θα τη βάλουμε και αυτήν μέσα. Αν δεν μας δώσουν εγγυήσεις, τότε νομίζω ότι ακολουθούμε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο. Δεν θα περάσει μόνο το 258 αλλά και το 273 και το 264 και το κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα πια με βάση το 40. Πολύ επικίνδυνος δρόμος λοιπόν. Τέλος. πρέπει να δούμε πώς θα βάλουμε την Κομισιόν σε κεντρική θέση σε αυτή τη συμφωνία. Αν τη δεχτούμε, γιατί φαίνεται ότι θα τη δεχτούμε, πώς θα βάλουμε την Κομισιόν στο κέντρο της, δίνοντάς της ρόλο σημαντικό και ρόλο κλειδί. Και πώς, πώς θα υπάρχει δημοκρατική λογοδοσία. How we can put Πώς μπορούμε να βάλουμε το κοινοβούλιο να παίξει το ρόλο του του πολιτικού ελέγχου. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον δικαστικό έλεγχο από το Ευρωδικαστήριο. Αυτά ήθελα να σας πω για αρχή. Ευχαριστώ και τους τρεις για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ο κύριος Ταρκόφσκι από την Επιτροπή ΑΦΚΟ ζητάει τον λόγο. Πρώτος. Δεν θα πω τίποτα καινοφανές. Κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαν οι παρατηρητές του Κοινοβουλίου. Για να συνοψίσω την θέση μας, όπως τη συζητήσαμε στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, έχω και ένα στοιχάκι, ότι η συνθήκη είναι πολύ μα, μακρός και λύσεων, θα πρέπει να είναι πολύ λιτή και είναι πολύ γενικόλογη, γιατί θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, μιλάει για όλα τα μέτρα που θα, που θα έπρεπε, ενώ πολλοί από εμά συμφωνούμε ότι αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να περάσουν μέσω ε, δευτερογενούς νομοθεσίας. Και είναι πολύ γενικό, λέγει, ό,τι αφορά το ρόλο των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή της ο Έλμαρ είπε για δύο πράγματα που είναι σημαντικά και άλλοι όμως τα έθιξαν ότι αυτή η συνθήκη θα πρέπει να είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και στα συμπεράσματα της Συνόδου είχε μπει αυτό το σημείο ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα σαφή ορισμό ότι αυτή η συνθήκη θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κάποια στιγμή να δημιουργηθεί η δυνατότητα να γίνει τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Αν συμφωνούμε ότι πολλά μπορούν να γίνουν από, μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας, ο στόχος μας θα πρέπει ε, να είναι, μια πολύ ε, λακωνική συνθήκη χωρίς όλες αυτές τις διατάξεις. Αν αποφασίσουμε για συμβολικούς λόγους ότι θα είναι πιο ευρεία, τουλάχιστον να έχουμε μια ρήτρα που να λέει ότι με την επιφύλαξη της δευτερογενούς νομοθεσίας μπορούν να γίνουν τα κάτωφη. Και επίσης ε, θεσμικό, ισχυρό θεσμικό ρόλο των κοινοτικών μας οργάνων ε, και για το άρθρο 273 ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχω τις αμφιβολίες μου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 273 ε, για το δικαστήριο. Έχω αμφιβολίες όπως είπε και ο Γουαλτιέρη Επίσης ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να γίνει, ε, θα πρέπει να γίνει με την επιφύλαξη του άρθρου 121. Το άρθρο 12 που το ανέφεραν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, που θέτει τα εθνικά κοινοβούλια όχι σε ίση βάση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τα προνόμια μας ε, με βάση αυτά τα άρθρα. Επίσης, για αυτά τα νέα όργανα, ε, ο τίτλος 5, προβληματικός. Γιατί αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την κοινοτική μέθοδο, δεν είμαι σίγουρος ότι χρειαζόμαστε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που να μιλάει για την ε, Σύνοδο Κορυφής κτλ. Τα έχουμε ούτως ή άλλως όλα αυτά στα συμπεράσματα τη Συνόδου προηγουμένω. Και τίποτα δεν υπάρχει να εμποδίσουν τα κράτη-μέλη να κάνω ό,τι πρέπει, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό βασικό τμήμα τη διακυβερνητική συνθήκη. Ε, πιο λακωνική συνθήκη, όπως είπα τελικά, αυτό είναι το βασικό, πολύ πιο συνοπτική, αλλά πολύ πιο συγκεκριμένη ό,τι αφορά το ρόλο των ε, οργάνων μας, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτά. Από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σώπα κορεδέ, σα ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να είμαι απλοϊκό. Εγώ ασχολήθηκα με το δίκαιο όλη μου τη ζωή, αλλά θα ξεχάσω ότι είμαι ε, ε και θα σα θυμηθώ ότι είμαι δήμαρχος με τους κλείσεις πόλεις 3.000 κατοίκων. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ποιότητα αυτού του εγγράφου. Δηλαδή, αν εργαστούμε πάνω σε κάτι ουσιαστικό, ή αν είναι κάτι το πολύ ασαφές που μας αποστέλλεται για να μπορέσουμε ε, να εργαστούμε με τη βεά μας ουσία. Δεύτερον, δεν θα πρέπει οι Βρυξέλλες να γίνουν Βαβυλώνα και όταν υπάρχει παντού κρίση εμείς ασχολούμεθα με κάποιες λεπτομέρειες νομικής μορφής που δεν ενδιαφέρουν κανένα. Δεύτερον, ρεαλισμός. Έδωσα μια ματιά στο κείμενο και λέω Μα τι είναι αυτό. Αν πάρουμε κατά λέξη αυτά που έχουν γραφτεί, που παντού αναφέρονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέω, ε, λοιπόν τότε τι, αυτή η συνθήκη είναι για να ικανοποιηθούν οι πολιτικοί. Διακοσμητικό είναι δηλαδή αυτό, όπως λέμε οι δικηγόροι. Και τότε ε, πώς θα το εξετάσουμε σαν είναι αναπόσπαστο μέρος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει έτσι να το προσεγγίσουμε για να δούμε τι θέλουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών. Κατά πόσον το έγγραφο που έχουμε έχει ουσία, κατά πόσον η στάση που έχουμε εμείς θα πρέπει να μην επεξηγεί τίποτα, αλλά να το πάρει κατά λέξη, να το πάρει κατά λέξη αυτό το κείμενο και σήμερα το απόγευμα κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα, ένα δημοσιογράφος που μου έλεγε «Η δημοκρατία επιβάλλεται, δεν συζητιέται. Ας αποδείξουμε ότι και το κοινοβούλιο μπορεί να επιβληθεί σε αυτή τη συζήτηση». Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή ΑΦΚΟ, ο κύριος Γκουερέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι η πρωτοβουλία που πήραν τα κράτη-μέλη και η οδός που ακολουθούν δεν προσφέρει ένα θεσμικό ρόλο στο Κοινοβούλιο. Τη στιγμή αυτή που διαπραγματευόμαστε αυτή τη διεθνή συνθήκη να δεχτούμε την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου ε, διαλέγοντας τρία άτομα που θα ενταχθούν ε, σε αυτή την ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της Κομισιόν και του, Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου. Ο ρόλος λοιπόν και η δύναμη του Κοινοβουλίου Ε, θα ενισχυθεί μόνο αν έχουμε εσωτερική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή ούτω ή άλλω είμαστε στο περιθώριο. Θα πρέπει εμεί να μιλήσουμε με μία φωνή, να έχουμε ενότητα. Ε, θα πρέπει να του πούμε τι πρέπει να υπερασπιστούν σε αυτή τη διαπραγματευτική προσπάθεια. Αν αρχίσουμε να συζητάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τουλάχιστον να καταλήξουμε. Αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να έχουμε συμφωνία των πολιτικών ομάδων. Γιατί αν δεν υπάρχει ε, συμφωνία των πολιτικών ομάδων ε, θα διαβρωθεί η ισχύ μας. Καταρχάς οι τρεις συμφώνησαν πάνω στην, στο όραμα και στη θεώρηση που πρέπει να έχουμε. Και συμφωνούν πώς, ε, ως προς το πώς θα επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αμφιβολίες θα πρέπει να τις ρυθμίσουμε. Ας πούμε, αν αυξήσουμε το περιεχόμενο της συνθήκης, αν επιλέξουμε αυτή την άγουσα, περνώντας μέσα από ένα άρθρο, το οποίο ε, εκ των υστέρων θα μπει στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν βάλουμε αυτή τη ρήτρα, τη sunset clause, που θα μας εγγυάται ότι τελικά τα βάζουμε όλα αυτά στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε στην πραγματικότητα αυξάνουμε το περιεχόμενο της σημερινής συνθήκης. Αυτό θέλουμε. Εάν πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια ε, θα πρέπει να συνθήσουμε αυτή τη διεθνή συνθήκη, η οποία θα υπάρχει παράλληλα με τις άλλες συνθήκες, τουλάχιστον να, το ξεκαθαρίσουμε αυτό το ερωτηματικό, τι θέλουμε και να πιέσουμε για αυτό που θέλουμε. Ορισμένοι μίλησαν για το περιεχόμενο που είναι κατώτερο από τη δευτερογενή νομοθεσία που υιοθετείται από το Κοινοβούλιο. Πέρα από αυτό το μικρό περιεχόμενο, έχουμε διάφορες άλλες αμφιβολίες. Δεν έχουμε δεν είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα αυτής της συμφωνίας, η οποία θα λειτουργεί με επικυρώσεις. Υπάρχουν χώρες που θέλουν αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν την έχουν επικυρώσει. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαιρέσεις και μεταξύ των κρατών μελών που θα υιοθετήσουν τη συνθήκη, αλλά που δεν, θα την, που δεν την έχουν υιοθετήσει, μάλλον δεν την έχουν επικυρώσει. Υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει διαδικασία μεταρρύθμισης. Εδώ επανερχόμαστε στη ρήτρα ηλιοβασιλέματος, αυτή τη sunset clause. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία τελικά δεν είναι πολύ ρεαλιστικά. Αν πιστεύουμε ότι αυτή η διεθνής συμφωνία πρέπει να μπει στην ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καθυστερήσουμε. Δεν θα ε, έχουμε γρήγορα στα χέρια μας τα οικονομικά στοιχεία που χρειαζόμαστε. Έχουμε επίσης την εντύπωση ότι ο στόχος αυτής της ε, πρωτοβουλίας είναι το να καταστήσουμε υποχρεωτικό το χρυσό κανόνα για το έλλειμμα για τις χώρες που ανήκουν στη ζώνη ευρώ και που θέλουν αυτή τη συμφωνία. Αλλιώς θα μπορούσαμε να περάσουμε μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία. Ή όπως προτάθηκε θα μπορούσαμε να είχαμε τροποποιήσει το πρωτόκολλο 12 για την ε, παρέμβαση που υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα. Σε περίπτωση που υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα. Η, η εφαρμογή του χρυσού κανόνα ε, είναι υπερβολικά έντονη Επίσης, μιλάμε για τη λεγόμενη ε, ισοδύναμη νομοθεσία ως προς, ως προς ένα σύνταγμα. Τι θα πει αυτό. Αν θέλετε να εμποδίσουμε το να, υπάρχουν προβλήματα επικύρωσης για χώρες που δεν θέλουν την τροποποίηση, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την λεγόμενη ισοδύναμη νομοθεσία. Αλλά ούτως ή άλλως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτή η ισοδύναμη νομοθεσία σε 26 χώρες. Αυτό μπορεί να σημαίνει από χώρα σε χώρα κάτι τελείω διαφορετικό. Ευχαριστώ, Ούτο Πούλμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που ανέλαβαν το τόσο σημαντικό αυτό έργο εξ το όλου του Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, κάθε τύχη που προσπαθείτε πραγματικά να προχωρήσει το θέμα αυτό εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκράτων στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Θα συνεργαστούμε, έχω να πω ότι θα συνεργαστούμε μαζί σα, θα σα υποστηρίξουμε, γιατί σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση είναι σημαντικό να δούμε τι δίνεται σαν απάντηση στην κρίση και πώς θα ενταχθεί αυτό στο κοινωτικό δίκαιο. Έχω όμως και δύο ερωτήσεις και ίσως κάποιες προτάσεις. Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα όταν λέγεται ότι οποιαδήποτε αντίδραση αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή της τελευταίας ε, συνόδου κορυφής θα πρέπει να ενταχθεί στην κοινοτική μέθοδο να αναφερθεί στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί συνήθως ε, υπάρχει πρόταση της Κομισιόν και δύο συν νομοθέτες, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που συμφωνούν κάπου. Αυτό έγινε και με το Six Pack, ε, το λεγόμενο. Δεν είναι θέμα κατά πόσο μα αρέσει ή δεν μα αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά η δημοκρατική διαδικασία προβλέπει ότι συνεργάζονται τα δύο σώματα και καταλήγουν σε μία λύση την οποία ε, πρέπει πραγματικά να προασπίσουν και και να βελτιώσουν. Υπάρχουν στοιχεία που μου αρέσουν, υπάρχουν στοιχεία που δεν μου αρέσουν, αλλά είμαι τώρα πια υπεύθυνο γι' αυτό. Αυτή η μεταφορά μιας απόφασης των κρατών μελών μια διακρατική συμφωνία δηλαδή πώς θα περάσει στην κοινοτική νομοθεσία εάν εκ των προτέρων είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι δηλαδή πρόταση Κομισιόν, αλλά ο συνομοθέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο λέει ότι ναι, υπάρχει το αποτέλεσμα και εμείς μεθοδικά και μεθοδολογικά θα υιοθετήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι προβληματική η κατάσταση. ίσως θα ήταν καλό το αποτέλεσμα να είναι πιο ανοιχτό για μια νέα δομή. Γιατί αλλιώς δεν είναι αποτέλεσμα της κοινοτικής μεθόδου και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να υπάρχει στην ημερησία διάταξη των διαπραγματεύσεών μας. Και τώρα περνάω σε ένα άλλο σημείο, όπου έχω μια άποψη, αλλά θα κάνω και μια πρακτική πρόταση. Δηλαδή, Εάν ο πυρήνας της πρώτης των κρατών είναι η ε, δημοσιονομική ένωση, η χρηματοπιστωτική ένωση να είναι ένας αυτοματισμός, να μην εξαρτάται από αποφάσεις, να μην εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση, αλλά να είναι ένας αυτοματισμός και έχουμε αφενός ρευστότητα και άλλε τέσσερι εβδομάδε υπάρχει μια συνάντηση σε κρατικό, διακρατικό επίπεδο και λέμε τι γίνεται με την ανεργία, αυξάνεται και η, πώς προχωρά το θέμα με την οικονομική ανάπτυξη. Από τη μια στιγμή η φορολογική λιτότητα και από την άλλη μεριά συζητήσεις ε, μη δεσμευτικέ για τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τότε αυτή η συμφωνία δεν θα επιζήσει τις κρίσεις άσχετα το τι θα ψηφίσουμε εμείς εδώ στο σώμα, η εξέλιξη των αγορών, η εξέλιξη πραγματικής οικονομίας θα καταδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατακαιρματιστεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη, πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία, πώς θα ενσωματωθεί σε αυτό το κείμενο. Αυτή η μακροοικονομική διάσταση δηλαδή που υπάρχει και στην πρόταση της Κομισιόν για το λεγόμενο six-pack. Δεν σας λέω ότι θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή, αλλά θα πρέπει να απαντήσουμε το γενικό ερώτημα. Νομίζω ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις για το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο αυτό που αποφασίστηκε. Εγώ είμαι υπέρ της ε, δημοσιονομικής παγίωσης οπωσδήποτε. Αλλά τώρα πώς θα γίνει αυτό, αν δεν χρειάζεται και ανάπτυξη ταυτόχρονα, θα πρέπει να το δούμε. Αλλά αυτές οι ιδέες να τις δώσω στους τρεις συναδέλφους, να έχουν δηλαδή μια γενική εικόνα, αναγνωρισμένα ε, Ινστιτούτα ε, Οικονομικής Έρευνας ε, από το κύριο παραδείγματος χάρη αυτό, το Ινστιτούτο ή και άλλα Ινστιτούτα, ποιες είναι οι οικονομικές προγνώσεις που κάνουν βάσει αυτής της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης. Πώς διαβλέπουν την οικονομική εξέλιξη εάν γίνει αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Ίσως ε, τα στοιχεία αυτά να βοηθήσουν τους συναδέλφους να προωθήσουν τη συζήτηση. Με μια τέτοια πρόταση θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο άνετα πάνω στον πάγο στον οποίο βρισκόμαστε. Ο κύριο Ντάφ έχει το λόγο τώρα. Ε, πρόεδρε, πρόεδροι και συνάδελφοι. Αντιμετωπίζουμε εδώ τη μεγαλύτερη ρήξη που έχουμε ποτέ γνωρίσει ως προς το σύνηθες κοινοτικό σύστημα. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολη στιγμή και ιδιαίτερα πλήττεται η αρχή ότι δεν πρέπει τα κράτη-μέλη να προσπαθούν να δρουν εκτός του κοινοτικού πλαισίου, του ενωσιακού πλαισίου όταν μπορούν να δράσουν εντός του. Και γιατί χρειάστηκε αυτή η ρήξη, γιατί πρόκειται για ρεαλιστική λύση αντιμετώπισης του Βρετανικού βέτο. Θα γνωρίζετε ότι εγώ είμαι κατά του Βρετανικού βέτο δεν θα το εξηγήσω καν, ούτε θα το δικαιολογήσω. Είναι όμως γεγονός και δεν έχει νόημα τώρα να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει απλή λύση για να αλλάξει η Βρετανία τη στάση της και να δεχτεί αλλαγή της συνθήκης που είχαν υπογράψει οι 27. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι καλό στοιχείο έχει αυτή η συμφωνία. Το καλύτερο τη στοιχείο είναι η ευέλιξία που προβλέπουν οι ρήτρε της. Αυτό πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και να βγάλουμε συμπέρασμα. Όταν θα συζητήσουμε, όταν θα έρθει η στιγμή να συζητήσουμε πραγματική αλλαγή των συνθήκων. Ως προτεραιότητα πρέπει να προστατέψουμε και να προωθήσουμε τον ρόλο της Κομισιόν χωρίς προσφυγή στο άρθρο 352 πρόκειται στην ουσία για μια συμφωνία κυρίων που λέει ότι όλοι οι συμβαλόμενοι πρέπει να φερθούν ως κύριοι και κυρίες. Εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία που εξέφρασαν προηγούμενοι ομιλητές ως προς το ρόλο του δικαστηρίου που θα μπορούσε να γίνει και υπερβολικός και φοβάμαι ότι θα, μειωθούν, θα μειωθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ερωτώ λοιπόν και τους τρεις σας. Τι είπε η Κομισιόν για όλα αυτά το απόγευμα. Θα ήθελα να μου το πείτε. Να μου πείτε ακόμη και καμιά φήμη για το τι είπε η Κομισιόν. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι, πάλι και για τους τρεις σας, συμφωνήσατε μεταξύ σας. Εκεί το απόγευμα. The next speaker uh, is Sylvie Goulard, though I wonder whether we should be having a short... Η Σιλβί Γκουρό. Μήπως κανένας από τους ηγητές θέλει ήδη να απαντήσει ή στο τέλος. Αν απαντήσετε τώρα θα λάβουμε υπόψη και την απάντησή σας οι επόμενοι ομιλητές. Θα λάβουν υπόψη. Ήταν πολύ δηλωτικέ οι εκφράσει των προσώπων των ε, βουλευτών. Γίνεται συζήτηση εκτό μικροφόρου. Εγώ έχω μια προσωπική εκτίμηση. Δεν ξέρω αν εκφράζω και του άλλου δύο εισηγητέ. Έχω την αίσθηση ότι η Κομισιόν δεν έχει κάνει ενδελεχή ανάλυση. Ε, πήρε θέση χωρίς να έχει κάνει ανάλυση. Μέχρι τη δεύτερη φορά όμως ε, μας υποστήριξε. Υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα άρθρο. Ότι αργότερα, δηλαδή μέσω αυτού του άρθρου, θα μπορεί όλο το, το οικοδόμημα αυτό να εντάσσεται στις υπάρχουσες συνθήκες. Σιλβί. Ευχαριστώ. Μια πρώτη παρατήρηση. Δεν νομίζω ότι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα το βράδυ είναι το Βρετανικό βέτο. Δεν πρέπει να λέμε παραμύθια. Ξαναδιαβάσετε την ε, ε, ομιλία της ε, κυρίας Μέρκελ στις 2 Νοεμβρίου 2010, την επόμενη ομιλία του Σαρκοζή, υπάρχει μια θέληση να παρακάμψουν την κοινωτική μέθοδο. Και όλοι εσείς, γιατί υπάρχουν και άλλοι συγγητές για το six-pack, για τα έξι αυτά νομοθετικά κείμενα, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε αυτή την εμπειρία ε, και στα πλαίσια της νομοθεσίας που διαπραγματεύομαι, στα πλαίσια της συναπόφασης. Πολλοί ήταν οι ιδρυτικοί πατέρες της συνθήκης Λισαβόνας που εν συνεχεία δεν δέχονται αυτό το κοινοβούλιο να παίζει πλήρως το ρόλο του. Θέλω να το πω αυτό, να το πω εισαγωγικά, να το ξέρουμε. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε αυτό που φτιάξαμε μέσα σε 60 χρόνια απέναντι σε ανθρώπους που θέλουν να το παρακάμψουν και να γλιτώσουν από αυτό. Δεύτερον, από την εμπειρία στη Γαλλία μάθαμε ότι όταν διαπραγματευόμαστε μία συνθήκη θα πρέπει να την επικυρώνουμε κιόλα και να σκεφτούμε το θέμα της επικύρωσης. Θέλω να σας θέσω το εξή ερώτημα. Ίσως είναι αφελές. Δεν είναι τόσο έτσι λεπτό και ψαγμένο αυτά που είπατε, να μην διαρωτηθείτε αν είστε συνυπεύθυνοι. Κάποια στιγμή αυτή η συνθήκη θα πρέπει να την πουλήσετε και θα την παρουσιάσουν ως την απάντηση της Ευρώπης. Επομένως, η βασική ερώτηση που μας απασχολεί είναι εμείς δεχόμαστε αυτόν τον τρόπο οικοδόμησης Ευρώπης. Θέλω να μπω σε δύο θέματα εδώ και να σας πω ξεκάθαρα ότι εγώ προσωπικά αυτό το κείμενο δεν το θέλω. Δεν το προσυπογράφω. Παρότι ανήκω σε πολύ φιλοευρωπαϊκά ρεύματα και τάσεις. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να το πουλήσω στους πολίτες, στους Γάλλους, στους ε, εκλογείς μου, ακόμα και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή μια Ευρώπη η οποία ε, συμπεριφέρεται έτσι σε δημοκρατικό επίπεδο και σε ε, οικονομικό επίπεδο. Οικονομικά καταρχάς. Κάναμε μια μάχη. Όλοι, βάζαμε σε διαφορετικά σημεία την έμφαση, αλλά νομίζω ότι στο six-pack ε, υπήρχε όλο αυτό το καινοτόμο τμήμα που έλεγε ότι η κατάσταση, η κρίση δηλαδή, δεν ήταν θέμα το προϊόν της έλλειψης της πειθαρχία. Ήταν και συνέπεια της ύπαρξης μακροοικονομικών ανισορροπιών. Δηλαδή είχε τρία επίπεδα. Το έλεγχο το δημοσιονομικό, την εποπτεία τη δημοσιονομική και θετικές πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ, υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης κτλ. Ίσως δεν είχαμε το τρίτο στοιχείο στο six pack, αλλά εδώ ουσιαστικά ε, επιστρέφουμε στην αφετηρία. Ξεκινάμε Ξεχνάμε αυτά που συνέβησαν στην Ιρλανδία, στην Ισπανία. Δεν μιλάω για ιδεολογία, μιλάω για την πραγματικότητα. Η κρίση δεν προκλήθηκε μόνο λόγω των δημοσιονομικών ισορροπιών. Έχει πιο περίπλοκες αιτίε. Και η οικονομική απάντηση που θα πρέπει να δώσουμε θα πρέπει να είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτή που ε, έχει συνθήκη που είναι μπροστά σας. Επαναλαμβάνω ότι το να είναι ε, ένας απλός ελεγκτής η Ευρώπη που ελέγχει απλώς την ε, πειθαρχία είναι λάθος, λάθος. Και το λέω γιατί είμαι η συγγήτρια που πολέμησε ενάντια στη Γαλλία για την αυτόματη εφαρμογή των κυρώσεων. Το θέμα δεν είναι ε, πειθαρχία ή ανάπτυξη. Το θέμα είναι πώς θα συνοδεύσουμε τις πολιτικές λιτότητες σε οποίες χρειαζόμαστε εκ των όνου και που μερικές χώρες μέχρι στιγμής δεν θέλουν να βάλουν στην δευτερεύουσα νομοθεσία, ε, αλλά που την, τα βάζουν έτσι πολύ ισχυρά στην πρώτον γεννή νομοθεσία, χωρίς να έχουμε το άλλο, το άλλο στοιχείο. Επομένως, οικονομικά υπάρχει μια ανισορροπία εδώ και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να πολεμήσουμε. Αν τελικά υπάρξει αυτή η συνθήκη. Θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν. Επίση υπάρχει και κάτι τερατώδε και το λέω και το τονίζω ε, στην επαναχώρηση που κάνουμε σε ό,τι αφορά το θέμα της δημοκρατίας το να βάλουμε αυτό το πακέτο Europlus που το διαπραγματεύτηκε το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο, που είχε ε, καθεστώς δήλωσης και να το βάλουμε στη συνθήκη χωρίς αυτή η συμφωνία, αυτό το pact, να αφορά τα κοινωνικά θέματα, τη φορολογία και την οικονομική πολιτική, χωρίς αυτή η συμφωνία να έχει συζητηθεί ποτέ, ούτε στα εθνικά κοινοβούλια, ούτε στο δικό μας κοινοβούλιο, είναι μία ε, ένα κόλεφο για τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να πούμε στου ε, εκλογεί η Ευρώπη, η δημοκρατία. Δεν συμφωνώ. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε και Ευρώπη και δημοκρατία. Ε, προσπαθήσαμε στο Six Pack να βάλουμε κανόνε. Αυτοί οι κύριοι του Συμβουλίου θα μπορούσαν να του λάβουν υπόψη, γιατί είχαμε συμφωνήσει για οικονομικό διάλογο, δημόσιο. Ούτω ή αυτό θέλανε. Αν θέλετε να κάνετε peer pressure, να πιέσετε του τους ομότιμούς σας, γιατί να μην δεχτούμε, σεβαστούμε αυτό που υπάρχει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, όταν υπάρχει πρόβλημα και η Ευρώπη δίνει συστάσει, να κάνουμε δημόσια συζήτηση και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτή τη χώρα, α πούμε, που στυλιτεύεται να εκφραστεί. Γιατί για του κανόνε τη κινητικότητα ε, τη εργασία, τη ε, σύνταξη, τη φορολογία να μην γίνει δημόσια συζήτηση. Γιατί να γίνεται μονίμω συζήτηση και κλεισμένο το θυρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Φτιάχνουμε ένα, ένα τέρα που δεν λογοδοτεί σε κανένα που δεν έχει εκλεγεί ποτέ και που δεν δουλεύει δημόσια. Εγώ δεν βλέπω έτσι την Ευρώπη. Τελευταίο θέμα, τελευταίο ζήτημα. Υπάρχει ένα Κινέζο επενδυτή ή Αμερικάνο επενδυτή που μόλι διαβάσει αυτή τη συνθήκη θα πει: Α, ωραία να έρθουν επενδύσει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τέλεια. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, ο κύριος Έφνερ. Όταν τελειώσουν οι εισηγητές, οι συντονιστές συγγνώμη, να τοποθετηθούν οι τρεις εισηγητές μας, οι τρεις παρατηρητές του Κοινοβουλίου. Έτσι. Να τελειώσουν πρώτα όμως οι συντονιστές. Χέφνερ. Dank. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να διασώσουμε το ευρώ, καταστρέφοντας όμως την Ένωση. Αυτός είναι ένα κίνδυνος που πρέπει να έχουμε κατά νου. Γιατί θα, το τίμημα αυτό θα ήταν ε, απαράδεκτο. Και γι' αυτό και θέλω να πω εισαγωγικά πρώτα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ έτσι ενωμένοι και αυτό είναι κοινοβούλιο να μην συνεχίσουμε τα όπως τα πεπατημένα αλλά έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτε μέτρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω το άκουσα και από κάποιες παρατηρήσεις προηγουμένως για εμά που ασχολούμαστε με τα συνταγματικά θέματα, είναι σημαντικό λέω να εξάσουμε και οικονομικά θέματα και όχι μόνο να κοιτάμε πάντα την νομική πτυχή αλλά να εξτάσουμε και την οικονομική πτυχή και τα ναπαλίν. Το κοινοβούλιο στο σύνολό του θα πρέπει να εμπλακεί πολύ πιο ενεργά στη συζήτηση αυτή από ό,τι το είχε κάνει στο παρελθόν. Δεν θέλω να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για το εξή. Ε, αποφασίσαμε να οικοδομήσουμε αυτό το κοινό οίκο Ευρώπη. Και ίσως θα πρέπει να βασίζεται στο δίκαιο, στη δημοκρατία, στα θεμέλια ενό κοινού συντάγματο υπό τη μορφή μια συνθήκη. Και τι έχουμε τώρα. Δίπλα χτίζεται ένα αυθαίρετο που μπορεί κανένα να το ανοιχτεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα πρέπει η Ευρώπη στο τέλος να είναι ένα συνοθήλευμα αυθαιρέτων χωρίς πραγματική νομική βάση, αλλά θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό δίκαιο και στη δημοκρατία. Και θα ήθελα να πω στο τέλος αυτό που αναφέρθηκε όταν πρόκειται για το δημοσιομικό δίκαιο, το κεντρικό σημείο αυτών που διαβλέπουν οι πολίτες σαν νομοποίηση των κοινοβουλίων, σαν ε, το κύριο έργο ελέγχου των κοινοβουλίων, βλέπουμε τώρα ότι δίνεται ε, μεγάλη ισχύ, μεγάλη αρμοδιότητα σε κάποιο σώμα το οποίο δεν είναι ε, δημοκρατικά νόμιμο κατά κάποιο τρόπο. Και ακριβώς το θέμα της δημοκρατίας είναι το θέμα το σημερινό. Θα τα καταφέρουμε. Αυτό ισχύει και για τις ε, οικονομικές αγορές και λοιπά. Θα τα καταφέρουμε, λέω, η δημοκρατία να αποδειχθεί με αποφάσεις που τις επομίζονται και οι πολίτες να λύσει τα σημαντικά προβλήματα της σήμερον ή θα υποκύψουμε όλοι σε κάποιο ε, διευθυντήριο που αποφασίζει αυτά που μας αφορούν. Αυτό είναι πάρα πολύ ενσυγητικό, γιατί προσεχώς θα έχουμε κάποιες πάρα πολύ σοβαρές και αποφασιστικές ε, αποφάσεις να αντιμετωπίσουμε και αν δεν συζητηθούν και ελεγχθούν αυτές δημοκρατικά, τότε η Ευρώπη θα, αρχι, θα μπει σε, έναν, ε, ε, σε μια δίνη που θα την τραβήξει προς τα κάτω και όπου θα χαθεί η δημοκρατία. Αυτά εισαγωγικά. Δεν θέλω να πω τίποτα πάνω στην συνθήκη που έχουμε μπροστά μα. Τα είπα αυτά σήμερα τα απόγευμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Εγώ θέλω να υποβάλω κάποιες ερωτήσει στους αντιπροσώπους μα στην ομάδα αυτή εργασίας. Παραδείγματο χάρη, εμένα θα με ενδιαφέρε τις προσεκτική εβδομάδα. Πώ βλέπετε την, το συσχετισμό μεταξύ ε, ημών που είσαστε για μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό στην Τράπεζα των Επραγματεύσεων και τα διάφορα όργανα του Κοινοβουλίου. Δεύτερη ερώτηση. Ποιες είναι οι δυνατότητες που διαβλέπετε εσείς ρεαλιστικά το Κοινοβούλιο να μπορέσει να βελτιώσει το κείμενο ε, στο πνεύμα του δημοκρατικού ελέγχου και της κοινοτικής μεθόδου. Και επίσης, αν κατάλαβα αυτά που είπε ο Έλμαρ Μπρόκ, σωστά, είπε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που ζητούμε αυτό να τοποθετηθεί στην βάση του κοινοτικού δικαίου. Είπατε μάλιστα ότι υπάρχει πρόθεση αυτή η συνθήκη να περάσει στην κοινοτική συνθήκη προσεχώς. Και θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς μπορεί να γίνει αυτό, τι διαβλέπετε και σε ποια χρονικά διαστήματα. Ελπίζω ο Έλμαρ Μπρόκ να με ακούσει και να μπορέσει να μου απαντήσει. Μπορεί, μπορεί, ναι. Ακούει και, ακούει και μιλάει, δεν έχει σημασία. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα και τα δύο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ποιο θα μπορούσε να είναι το σεμινάριο βάσει το οποίο θα περάσει αυτό στην γενοτική μέθοδο. Με συνέλευση ή με δυναμωμένη συνεργασία ή πώς. Και επίσης ε, ποια θα είναι τα χρονικά διαστήματα που έχουμε εδώ κατά νου. Επίσης, η λεγόμενη sunset clause, η ρήτρα του ηλιοβασιλέματος. Πολύ ωραία ιδέα. Είναι ρεαλιστική όμως η ιδέα αυτή. Είναι ρεαλιστική αυτή η συνθήκη να έχει ένα, μια ρήτρα ε, Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές όταν πούμε αυτό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, ε, Φερρυπίν. Εγώ δεν φαντάζομαι να είναι πολύ ευτυχεί οι αγορέ. Λέει ο πρόεδρο. Επόμενο ομιλητή. Okay, ich werde auch mal Deutsch sprechen hier. Να μιλήσω κι εγώ γερμανικά, έτσι. Λοιπόν, μου είπαν ότι ο Έλβαν Μπρουκ μπορεί και να ακούει και να είναι multitasking παρόλο που λένε ότι το δικό μας το φίλο δεν ειδικεύεται στο να ασχολείται με πέντε πράγματα ταυτόχρονα. Λοιπόν, ε, ο κίνδυνος ε, αναφέρθηκε ότι ε, μπορεί να σώσουμε το ευρώ και να θάψουμε την Ένωση, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνο αυτό γιατί αυτή η συνθήκη δεν πρόκειται να σώσει το ευρώ. Δεν επιτρέπεται να ε, κάνουμε εδώ ένα διπλό σφάλμα. Και εάν στην σημερινή παγκόσμια οικονομική κατάσταση τραβήξουμε τα ενία τόσο πολύ, ξέρουμε ότι ταυτόχρονα το μόνο που δεν θα καταφέρουμε είναι η εξυγίαση των προϋπολογισμών των κρατών. Γι' αυτό θα υπάρχει λοιπόν οικονομική αποτυχία εάν δεν υπάρχουν ταυτόχρονα διορθωτικά μέτρα που θα μπορέσουν να δώσουν κάποια εκτατικ... κάποιες εκτατικές οθήσεις. Και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να μιλάμε για δημοσιονομική ένωση, όπως λέγεται συχνά, γιατί αυτό θα συμπεριλάμβανε ένα τμήμα της εξυγίασης των προϋπολογισμών, αλλά θα έχει και κανόνες όσον αφορά τα έσοδα, δηλαδή τη φορολογία, και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κρατών μέσω των αγορών. Σήμερα και χάσει τη συνεργασία της Ελβικουλάρ, είπαμε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ότι χρειάζομαστε να υπάρχει κάποια μορφή ευρωομολόγων με αυστηρούς κανόνες. Και αυτό λείπει και ξέρουμε γιατί λείπει, γιατί υπάρχουν ακριβώ αντιδράσει σε εκείνη τη συγκεκριμένη χώρα, χάρη τη οποία έχουμε όλη αυτό, αυτή τη συνθήκη. Αυτή τη χώρα που και εγώ καλύτερα γνωρίζω από οποιονδήποτε. Άρα αυτή, αυτή η συνθήκη που προτείνεται δεν είναι μια σωστή απάντηση προς την κρίση και έτσι το βλέπουν και οι αγορές. Τα spread δεν μειώθηκαν σημαντικά, τουλάχιστον όχι μακροπρόθεσμα. Γιατί η Κεντρική Τράπεζα άνοιξε την, ε, τη ροή του χρήματος και γι' αυτό βλέπουμε σε ορισμένε χώρες μείωση των spreads, βραχυπρόθεσμα όμως, όχι μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα μηνύματα να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς ως πολίτες και ως εκλεγμένοι από τους πολίτες πάρουμε σοβαρά υπόψη την εντολή μας, θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να κάτσουμε σαν παρακαθήμενοι σε αυτή τις διαπραγματεύσεις και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια βελτίωση. Και σας ευγνωμονώ βέβαια για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε, αλλά δεν μπορεί αυτή να είναι η μόνη αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε αυτή τη μονομερή προσπάθεια αντίδρασης στην κρίση. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, εκ με τις προσπάθειες για τη λεγόμενη δημοσιονομική συμμαχία, εκ παραλίλου λέω να υποβάλλουμε δικές μας προτάσεις ως Κοινοβούλιο εκ παραλίλου με τον ίδιο ενθουσιασμό με τον οποίο συμμετέχουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή είναι σωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβάλει δικές του προτάσεις σε αυτή την, ε, αυτή την ομάδα εργασία, αποφάσισε και η διάσκεψη των Προέδρων, αλλά, και θα πρέπει να το πούμε αυτό στι συγκεκριμένε διαπραγματεύσει, εάν δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό, αυτή η συμφωνία θα αποτύχει και δεν θα πρέπει εμείς να δώσουμε την ευρωπαϊκή μας ευλογία ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Εάν το κάνουμε, δικαίως θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας αργότερα για μια αποτυχία. Σας παρακαλώ, συζητήστε με τους οικονομικούς σας συμβούλους και συζητήστε με οικονομικούς συμβούλους διαφορετικών προελεύσεων. Και ο συνάδελφος Μπούλμαν το ανέφερε προηγουμένως στο Ινστιτούτο για την διεθνή οικονομία στο Κίελο, που οπωσδήποτε δεν είναι αριστερό, είπε ότι οι απαιτήσει αυτή τη ε, δημοσιονομικής συμφωνίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γιατί τα απαιτούνται θυσίες οι οποίες θα οδηγήσουν την ε, Ένωση σε ύφεση. Εγώ ξέρετε ήμουν πάντα υπέρ τη δημοσιονομικής πειθαρχίας. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Αλλά η μονομερή συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από τα νομικά. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως υπάρχουν και νομικά προβλήματα και επιχειρήματα, γιατί θα πρέπει εμείς ως Κοινοβούλιο να γνωρίζουμε ακριβώς τα νομικά μας επιχειρήματα, παραδείγματος χάρη. Μέσω της πρώτη αυτής ε, μήπως καταπατέται το δικαίωμα πρωτοβουλία της Κομισιόν σε τομείς που αφορούν την ε, κοινοτική πολιτική. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορές μεταξύ του six και αυτού του λεγόμενου ε, κειμένου δημοσιονομική ε, ε Αναφέρει και ο κύριος Γκουλιέρη κάτι παρόμοιο. Και αν αυτά είναι αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα, έξω από τα δόντια. Και θα ήθελα επίσης να ξέρω τι σημαίνει ότι τώρα ένα τμήμα του six-pack γίνεται πιο αυστηρό όσον αφορά τη μορφή με την οποία εφαρμόζεται, το άλλο τμήμα του six-pack όχι. Αυτά είναι σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε αυτού του τύπου τα επιχειρήματα και να υποβάλουμε και δικές μας προτάσεις. Και, και τελειώνω, μια επίπτωση θα είναι επίσης, εάν εμείς αυτό το την παράλληλη συμφωνία δεν μπορούμε παραλίγο να αντιδράσουμε σαν κοινοβούλιο, θα πρέπει παρόλα αυτά να ξεκινήσουμε, να ζητήσουμε μία αλλαγή της συνθήκη εμείς, ούτως ώστε να περάσει όλο το θέμα αυτόματα στην κοινοτική μέθοδο. Δεν μπορεί κανένας να μας απαγορεύσει να ζητήσουμε να υπάρχει μία συνέλευση και οι περισσότεροι πολίτες θα είναι οπωσδήποτε στο πλευρό μας όταν προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως Βρετανός που παρακολουθεί τις εξελίξεις θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Πρώτον, τη προφανής. Δεν πρόκειται για ενωσιακή συνθήκη και άρα το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παίξει επίσημο θεσμικό ρόλο. Σίγουρα το Συμβούλιο θα ακούσει πολύ ευγενώς αυτά που μας είπαν οι τρεις μας σοφοί. Θα ακούσει ό,τι έχουμε να πούμε και μετά θα συνεχίσει να κάνει οτιδήποτε είχε σκοπό να κάνει. Διότι παρά το ότι το Βρετανικό βέτο το πρόσεξαν πολύ, αυτό έκρυψε, απέκρυψε το γεγονός ότι πολλές χώρες μέλη δέχονται μια διακυβερνητική συμφωνία, είναι ικανοποιημένε. Θα με εξέπλησε πολύ, μπορώ να, κάνω και, να βάλω και στοίχημα με τον κύριο Φερχόφσταντ, αν και οι 26 χώρες δεχόνταν, δέχονταν αυτή τη συνθήκη. Αυτή η νέα λοιπόν δομή δεν είναι καθόλου θεμητή ούτε νόμιμη. Το έχουν, με την έχουν μεν δεχτεί εθνικές κυβερνήσεις που είναι υπόλογες στα εθνικά κοινοβούλια και εδώ αυταπατώμεθα νομίζουμε ότι είμαστε το μόνο όργανο που εγγυάται τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Εγώ συμφωνώ με πολλά από αυτά που λέει ο Ζαν Πολ Γκοζές. Γιατί ο πειρασμός τέτοιων συναντήσεων είναι να δαπανάμε πολλή ενέργεια για νομικά κείμενα που καταφέρνουν πολύ λίγα πράγματα. Οτιδήποτε και να πούμε σήμερα δεν θα λύσει την κρίση. Είτε πρόκειτο για συμφωνία των 27 ή των 26 ή και λιγότερον. δεν θα άλλαζε αυτό τίποτα ως προς την τύχη της Ένωσης και του Ευρού. Γι' αυτό εδώ κάνουμε δραστηριότητες απόκρυψης στην ουσία, προπετάσματος καπνού. Αντί να συζητάμε αυτά τα πράγματα, ας συζητήσουμε τη θεσμική αλλαγή. Ας φανταστούμε ότι σε έξι μήνες περνάει αυτή η συνθήκη, ποια θα ήταν τα αποτελέσματά της ίσως να απέτρεπε την επόμενη κρίση σε 5 ή 10 χρόνια, αλλά δεν θα είχε καμία απολύτως επίπτωση επί της τύχης του ευρώ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ευρώ είναι πρόβλημα της αρχικής του σύλληψης. Δηλαδή, βάλαμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, επιβάλαμε στις χώρες μέλη που δεν μπορεί καμία να τα λύσει, ναι. Το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν υπερβολικό χρέος, αλλά αν η καγκελαρία Μέρκελ είχε ένα μαγικό ραβδί για να εξαφανίσει το χρέος αυτό, θα βλέπαμε ότι σε 10-20 χρόνια το ίδιο πρόβλημα θα εμφανιζόταν πάλι. Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι πολύ άκαμπτες οι αγορές εργασίας, πολύ ψηλοί οι φόροι και ο δημόσιος τομέας πολύ μεγάλος. Η Γερμανία κάθε χρόνο κερδίζει ένα ή εκατο μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα όσο υπάρχει το ευρώ, ενώ παράλληλα ένα με εκατο αποτελεσματικότητος χάνουν οι υπόλοιπες χώρες. Και αυτό οφείλεται στο ευρώ. Αν είχαμε κανονική φορολογική ένωση, αν ήθελε η Γερμανία να δώσει 10% του ΑΕΠ στις χώρες του Νότου, δηλαδή μια σταθερή επιχορήγηση, μπορεί να δούλευε το πράγμα, αλλά δεν βλέπω να θέλει τίποτα τέτοιο να κάνει η Γερμανία και δεν, τους, δεν το θεωρώ παράλογο αυτό, ούτε η χώρα μου θα το έκανε. Το πρόβλημα λοιπόν όπως το βλέπω εγώ είναι ότι μιλάμε όλοι για λάθος θέμα. Θα έπρεπε να μιλάμε για το πώς χώρες σαν την Ελλάδα και την Πορτογαλία θα επανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Και αντί γι' αυτό μιλάμε για αλλαγές των συνθήκων. Καλή τύχη κύριε, αλλά φοβάμαι το χειρότερο. Thank you. Um, όπως και ο προταλής σας ε, και όπως φαντάζεστε, ε, είμαστε και οι δύο Βρετανοί, αλλά εγώ θα μιλήσω λιγάκι διαφορετικά. Οι τρεις ε, εισηγητές χρησιμοποίησαν διάφορους όρους για αυτή την πρόταση είπαν ότι αυτές οι αλλαγές γίνονται για πολιτικούς και συμβολικούς λόγους, μεταξύ άλλων. Ε, νομίζω ότι ακολουθείται μια πολύ επικίνδυνη άγουσα όμως. Όπως οι διάφοροι ξένοι επενδυτέ, αρχίσουν να καταλαβαίνουν ε, τα ωφέλη και τις επιπτώσεις του πακέτου της οικονομικής διακυβέρνησης και καθησυχάζονται, ε, Τώρα εμείς με αυτά που κάνουμε τους ε, αποπροσανατολίζουμε ξανανοίγοντας μια συζήτηση για το ίδιο πάλι θέμα, οικονομική διακυβέρνηση, με μόνο σκοπό να περάσουμε από την ε, δευτερογενή στην πρωτογενή νομοθεσία. Οι επενδυτές δεν θέλουν τέτοιες διαταραχές, θέλουν ασφάλεια. Δεν θέλουν άλλη ανασφάλεια, θέλουν ε, ηγεσία, θέλουν ανάπτυξη. Η διαφορά μεταξύ μιας αλλαγής της συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και δεν θα φέρει ε, παγκόσμια κεφάλαια στην Ευρωζώνη. Οι επενδυτέ είναι αυτοί που έχουν του τίτλου των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων. Ε, θα είναι οι μελλοντικοί αγοραστέ των μελλοντικών τίτλων. Και είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και των 27 κρατών μελών. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε προγράμματα μελλοντικά εστιάσουμε στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. Ε, αν τα κρατημέλη δεν εμπιστεύονται το ένα το άλλο για να εφαρμόσουν το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης που ξοδεύσαμε ένα χρόνο το διαπραγματευτούμε, αν δεν εμπιστεύονται τα μέντα, δε, γιατί τότε οι επενδυτές να μας εμπιστευτούν, να εμπιστευτούν οποιονδήποτε, όταν δεν υπάρχει ε, ούτε κανονισμός ούτε συνθήκη, η εμπιστοσύνη είναι το βασικό. Το βασικό είναι ότι κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν πια. Θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των επενδυτών, θα πρέπει να εμπιστευτούμε οι μεν τους δε, θα πρέπει οι αγορές να μας εμπιστευτούν. Οι εκλογές μου δεν καταλαβαίνουν καθόλου αυτή τη συζήτηση και τι θα επιφέρει η αλλαγή στη συνθήκη. Και πραγματικά και εγώ σας λέω δεν καταλαβαίνω γρή. Honorable Sondergaard, AFCO. από την ΑΦΚΟ. Έφυγε όμως. Δεν είναι εδώ. Γιώργαν Κρούτερ. Ja, ich möchte mal vorwegschicken, Ευχαριστώ. Εγώ έχω να πω ότι δεν συμμεριζόμαι με τον ευρωσκευισμό του Κάμερον, αλλά αναρωτιέμαι πως θα πρέπει να του είμαστε ευγνώμων που ως 27 ο αρνήθηκε να υπάρχει άμεσα μια αλλαγή της συνθήκης. Αν δεν είχε αρνηθεί θα είχαμε διαφορετική συζήτηση και θα είχαμε ε, ε, αυτή τη στιγμή ξεκινήσει την τροποποίηση της συνθήκης Λισαβόνας. Αυτή θα ήταν η ησυχία μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το αξιολογήσουμε διαφορετικά το ότι αρνήθηκε να υπογράψει παρόλο που ε, τους λόγους για τους οποίους το έκανε δεν το συμμερίζουμε. Πολλά ελέγχθησαν ήδη. Δεν θέλω κάποια στιγμή από αυτά να τα ε, υπογραμμίσω, ιδίω αυτό που είπε η Σιλβή. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου είναι κάτι που και εμένα με εντυπωσίασε σε όλες τις διαπραγματεύσεις που είχαμε ε, ως ε, ΕΚΟΝ πάντα το ε, Συμβούλιο προσπάθησε να πείσει το Κοινοβούλιο για τις απόψεις του ή και να το θέσει κατά μέρο. Δηλαδή το Συμβούλιο ή για να το πούμε ξεκάθαρα τα κράτη-μέλη, ενοχλούνται πάρα πολύ που το Κοινοβούλιο έχει διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση ε, που υποθάπτεται εδώ που το Κοινοβούλιο προσπαθούν να χάσει τα δικαιώματα που του δίνει στη θήκη του, της Λισαβόνας και θα πρέπει εμείς να τοποθετηθούμε σωστά, να απαιτήσουμε το ρόλο που μας αρμόζει. Επ' δεν μπορώ παρά να τονίσω αυτά που είπε και ο Σφεν Κίγκουλ προηγουμένως. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι κάνει αυτή η συνθήκη, γιατί παίρνει κάποιες Πτυχέ του Sixpack που τέθηκε σε ισχύ στις 13 ε, τρέχοντος μηνός και αναρωτιόμαστε γιατί εφόσον αυτό έχει τεθεί σε ισχύ ήδη θα πρέπει να το εντάξουμε και σε μια διακρατική συνθήκη. Και υπάρχουν και κάποιες ε, πτυχέ που αφορούν την ε, δημοσιονομική πειθαρχία, μπορούμε να πούμε. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά τι μακροοικονομικέ ε, ανισορροπίε, είναι αδύναμα μένει στο six αλλά υπάρχουν όμως και δεν χρειάζεται να τα αποδυναμώσουμε ακόμα περισσότερα εάν τονίσουμε την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε και να στηρίξουμε επί και ότι η, η Γερμανίδα Καγκελάριος είπε ότι τα Ευρωμπόντ δεν τα συζητάμε πια, παρόλο που το Κοινοβούλιο ξεκίνησε, ξεκίνησε εδώ κάτι για το προεπολισμό και για το six-pack και θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό οφείλεται στην Σίλβη, πρέπει να το, να το τονίσουμε. Αλλά το να πει ότι εντάξει τελείωσε πάει, ε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, είναι παράδεκτο τελείω. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι εκεί που θα πρέπει να επιμείνουμε είναι κάτι διαφορετικό, γιατί αφενός έχουμε την εσωτερική αγορά, από την άλλη μεριά συζητάμε για ε, λύματα εξωτερικού εμπορίου και πλεονάσματα εξωτερικού εμπορίου ενός κράτους μέλους. Είναι αυτό πολύ ενδιαφέρον γιατί καταδεικνύει τις διαρθρωτικές ελλείψεις της εσωτερικής αγορές Πιστεύω ότι και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή η βάση αυτών που υπάρχουν σε αυτή τη ε, διακυβερνητική συνθήκη. Και θα ήθελα επίση να τονίσω, μέχρι flashback, ο, που το ξέρετε, που είναι ο ε, επικεφαλής οικονομολόγος της UNCTAD, του Οικονομικού Τμήματος δηλαδή του Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πλιστάκης τόνισε ότι οι αιτίε για τα ελλείμματα και τα δημοσιονομικά ελλείμματα βρίσκονται κυρίως στις μακροοικονομικές ανισορροπίες και ότι κατά βάση ο στόχος του 2% πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και εκείνοι που βρίσκονται υψηλότερα πρέπει να μειώσουν, αλλά και εκείνοι που βρίσκονται χαμηλότερα, όπως η Γερμανία παραδείγματος θα πρέπει να προσεγγίσουν αυτό το 2% δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε απόλυτα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, αυτή η ιδέα, ένα επιχείρημα που μπορεί κανείς πραγματικά να το δεχθεί και δεν έχει ακουστεί καθόλου στην όλη συζήτηση. Και γι' αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλέσαντες ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, αντισταθούμε. Ευχαριστώ. τελευταίος Ο κύριος Ένιου. Είναι εδώ. Thank you, Chairman, but I Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι όμως συντονιστής. Στη Βρετανία έχουμε την έκφραση πίσω στις ρίζες. Και αυτό θα ήθελα να πω και σε αυτή τη συνεδρίαση. Τελευταία στιγμή μας φωνάξατε είναι σημαντική φαίνεται συνεδρίαση αν κρίνω από τους δημοσιογράφους που κυκλοφορούσαν εδώ και ένας ευρωβουλευτής, η κυρία Θήνη έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα λυπούμενη γιατί δεν μπορούσε να προσέλθει αν και προβλεπόταν αύριο συνεδρίαση της ΑΦΚΟ που όμως ακυρώθηκε και υπάρχουν πολλοί ακόμη που έφυγαν πρόωρα. Στη Βρετανία επίσης λέμε τον κόσμο τον κυβερνάνε όσοι ξυπνάνε νωρίτερα. Δεν είναι σωστό να φεύγουν πριν την ώρα τους οι συνάδελφοι και αυτή η επιστροφή στις ρίζες σημαίνει ότι δεν υπάρχει νέα συνθήκη ενωσιακή καινούρια μετά την τελευταία πριν από 10 χρόνια. και κάποιος άλλος συνάδελφος που ξεχνάω το όνομά του γιατί δεν μπορώ να το προφέρω ανέφερε δεκάδες άρθρα για να δικαιολογήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βέτο. Ε, τότε πώς υπήρξε. Διακυβερνητική διάσκεψη για το ευρώ δικαίωμά τους. Αλλά μπορεί να καταλήξει σε συμμαχία ορισμένων χωρών μόνο που μπορεί να δεχτούν να γίνουν και ενιαία χώρα γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σωθεί το ευρώ. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Από τους εθνικούς βουλευτάς θα αποφασιστεί αυτό και όχι από τους ευρωβουλευτάς. Δεν πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να τους επηρεάσουμε και να υποκατα... τους υποκαταστήσουμε. Η δουλειά των ευρωβουλευτών είναι πώς να αντιδράσει η Ένωση σε αυτήν ε, την διακυβερνητική. Η ιδέα ευρωπαϊκή δικαιοσύνη είναι το ποτηρητής των συνθήκων και όχι η διαμεσολαβητής για διάφορους ποδοσφαιριστάς. Τι ρήτρε των συνθήκων επιτρέπουν να γίνει με αυτόν τον τρόπο μια συνθήκη να χρησιμοποιηθεί δηλαδή εξοκινοτική μέθοδος. Ίσως ο κύριος Φερχόφστατ μπορεί να απαντήσει η νομική υπηρεσία είπε ότι επιτρέπεται κάτι τέτοιο και αν όχι τι συμπέρασμα βγαίνει αν αρνήθηκε να αποφανθεί μάλλον η νομική υπηρεσία και οι 27 χώρες μέλη έχουν δώσει τη συνένεσή τους δεν το ξέρω, ερωτώ έχει αξιολογηθεί πόσο κοστίζει για το φορολογούμενο και τη φορολογούμενη η διοργάνωση τέτοιων συμφωνιών Νομίζω ότι υπερβάλλεται κατά πολύ, ξεπερνάτε την εντολή μας όλοι και πρέπει να λήξει αμέσως αυτή η συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα οι απλοί ομιλητές και ομιλήτριες τελείωσαν οι συντονιστές. Πρώτα τα μέλη της εικόν. Uh, Αυτοί από την ΑΦΚΟ. Από την εικόνα, από την εικόνα. Την ΑΦΚΟ έχουμε. Η Γκουρμάη. Um, uh, uh, Μερικοί πρέπει να φύγουν, αλλά τέλος πάντων, Ελίζα, είσαι η πρώτη. Ευχαριστώ. Θέλω να σας εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε εσά τους τρεις που, είσαστε, που συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να υπενθυμίσω όμως ότι τελικά δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Είναι παρατηρητής, υποτίθεται. Τελικά θα προσυπογράψει το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω από αυτά που λέγονται. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν καθόλου ποια είναι η θέση μας. Τώρα, για το περιεχόμενο. Οι εξηγήσει των αιτίων της ε, κρίσης είναι τελείως λανθασμένες. τα ελλείμματα και το χρέος δεν είναι η αιτία, είναι συνέπεια των ανισορροπιών που αυξήθηκαν στην Ευρώπη. Οικονομικές ανισορροπίες καταρχήν, αλλά είναι και συνέπεια της έλλειψης οριμότητας κατά την οικοδόμηση του ενιαίου νομίσματος. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, τα οποία υπέβοσκαν ούτως ή άλλως και υπήρχαν και τη στιγμή που πήραμε την απόφαση για το six-pack. Με την κοινοτική μέθοδο στο Κοινοβούλιο οργανώσαμε αυτή την εξέταση. Η νομοθεσία υπάρχει. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, είναι, εξής, είναι το εξής. Τι προσθέτουμε σε μια νομοθεσία που υπάρχει ήδη. Όταν βλέπουμε τη σύνταξη του κειμένου αυτού, βλέπουμε ότι επιλέξαμε συγκεκριμένα πράγματα που προέρχονται από το six-pack. Αλλά όπως είπε και πολύ σωστά ο κ. Γκουαλτέρη, υπάρχουν και πράγματα που έχουν αλλοιωθεί εντελώ, έχουν αλλάξει εντελώ. Επομένως, σε τι μας εξυπηρετεί σε οικονομικό επίπεδο το να έχουμε ένα απόσπασμα από μια νομοθετική προσπάθεια που έχει γίνει βγάζουμε δηλαδή κάποια πράγματα και κρατάμε κάποια άλλα. Και τελικά το τελικό αποτέλεσμα έρχεται σε αντίφαση με το six pack. Υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Υπάρχουν, υπάρχει το θέμα της α, ανάπτυξης, των ευρωμολόγων, όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στο six pack και εδώ δεν υπάρχουν, εξαφανίστηκαν. Πού πήγαν? Έπειτα ένα άλλο θέμα, το θεσμικό θέμα, που προστίθεται, που είναι δίπλα στην κοινοτική μέθοδο. Σε τι, τι εξυπηρετεί η κοινοτική μέθοδος, σε τι εξυπηρετεί. Είναι περίπλοκη. Αλλά μόνο χάρη σε αυτή θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν ε, σεβόμαστε την κοινοτική μέθοδο, Ακολουθούμε τη διακυβερνητική μέθοδο, εξού και τα προβλήματα που δημιουργούμε. Μία διακυβερνητική η διαθεσμική, αν θέλετε, μέθοδος είναι περίπλοκη. Εμείς έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε μια μέθοδο που θα εξασφάλιζε την ισορροπία ανάμεσα στα ισχυρά και στα αδύναμα κράτη. Δεν μπορούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να παραμείνουμε παθητικοί θεατές απέναντι σε μια διαδικασία που αμφισβητεί όλη την κοινοτική ισορροπία. Και με βάση αυτή την ισορροπία εξάλλου οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, για μένα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ προβληματικά. Μετασχηματίζουμε τη συνθήκη ή μάλλον με, μετασχηματίζουμε σε συνθήκη μια ερμηνεία λανθασμένη και παράλληλα γινόμαστε συνένοχοι σε μια διαδικασία που πολιτικά και θεσμικά είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτικές καταστάσεις σε μια περίοδο όπου οι πολίτες περιμένουν πράγματα, περιμένουν απαντήσεις απτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντήσεις στην κρίση. Ευχαριστώ. μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διερωτώ με πως και άλλοι συνάδελφοι ε, για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Φυσικά και εγώ εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους τρεις ε, παρατηρητές. Αλλά χρειαζόμαστε μια συνθήκη για να δούμε πώς θα συντονίσουμε τις ε, δημοσιονομικές πολιτικές. Ενώ τη στιγμή που χρειαστήκαμε ένα χρόνο για να συζητήσουμε ξανά και ξανά όλα αυτά τα προβλήματα στα πλαίσια του six-pack. Διερωτώ με μήπως αυτή η διαδικασία ακυρώνει την ε, μακρά υπομονετική ε, δημοκρατική δουλειά που μας οδήγησε στην υιοθέτηση τελικά του six, του six pack. Όπως είπε ο κύριος ε, Γκερέρο Σαλόμ, αυτά που είπε μάλλον σωστά, το κείμενο που μας προτείνουν σκληραίνει πολύ περισσότερο το, σύμφωνο σταθερότητας, πολύ περισσότερο το six pack. Βάζει κυρώσεις που γίνονται αυτόματες, γιατί βάζει τον ε, κανόνα της αντεστραμμένης ειδική πλειοψηφίας που είχαμε απορρίψει στο six αλλά κυρίως επανέρχεται στην αρχή του 3%. Σας υπενθυμίζω ότι στο Six Pack είχαμε βάλει ένα αριθμό μείωσης του ελλείμματος, 1% του ΑΕΠ κατ' μέχρι να φτάσουμε στο 3%. Εδώ είμαστε κάτω από το 3%. Πάμε πέρα από τη συνθήκη του Μάστρικτ. Ε, βάζουμε το 0,5% του, του διαρθρωτικού α, ελλείμματος που γίνεται δογματικό είναι 0,5% του διαφθορτικού ελλείμματος μαζί με τους ε, τόκους που εξυπηρετούν το χρέος. Δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφθορτικό το έλλειμμα. Αυτό ε, είναι συμβατό με το 3%. Αλλά ένα έλλειμμα διαρθωτικό που βάζει και τα, τους τόκους εξυπηρέτησης του χρέους δεν συνάδει με το 3%. Αυτό τι σημαίνει, ότι βάζουμε μέτρα λιτότητας ύψους 2,5% του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες. Για να καταλάβετε καλά, μια χώρα όπως η Γαλλία έχουμε διαφθορτικό έλλειμμα 3%. Το διαφθορτικό έλλειμμα χωρίς τους στόκους είναι 0,5%. Βλέπετε τη διαφορά, 2,5%. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά λοιπόν. Να σου τονίσω επίσης ότι οι πολιτικές που προτείνονται σε αυτό το κείμενο υπήρχαν, ή μάλλον ήταν αυτές που μας οδηγούσαν στην ύφεση. Η Γαλλία, που είναι ένας από τους πυλώνες του, του σκληρού πυρήνα, έχει μπει σε ύφεση μόλις τώρα. Προσοχή λοιπόν, αυτό το σύμφωνο, ή μάλλον αυτή η συνθήκη για να το πω έτσι, δεν θα ρυθμίσει τίποτα, δεν θα λύσει τίποτα. Μάλιστα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει την αντίδραση των λαών μας, γιατί το να βάλουμε το χρυσό κανόνα σε ένα σύνταγμα θα γίνει για πρώτη φορά. Θα βάλουμε δηλαδή την αρχή της οικονομικής πολιτικής σε ένα συνταγματικό ε, κείμενο. Ε, σε πολλές χώρες για κάτι πολύ λιγότερο είχαν πει όχι σε μια συνταγματική συνθήκη. Έτσι, για πολύ λιγότερα μέτρα. Και επίσης, αν έπρεπε να τροποποιήσουμε τη συνθήκη, ε, όπως είπε και ο Ζαν Πολ σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει πραγματική συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το υποομοσπονδιακό επίπεδο που πολλοί από εμά υποστηρίζουμε. Ακόμα και αυτοί που, α, μην ξεχνάτε ότι αυτοί που δεν είναι φεντεραλιστέ δεν είναι τμήμα τη συζήτηση. Για να επιβάλλουμε το υποομοσπονδιακό επίπεδο, να επιβάλλουμε το, λόγο, το ρόλο τη κεντρική τράπεζα. Οι κεντρικοί μα διοικητέ δεν μπορούσαν να παρέμβουν, γιατί δεν του το επέτρεπε το καταστατικό τη κεντρική τράπεζα. Ενώ τώρα ήγηκε η ώρα για να παρέμβουν. Θα μπορούσαμε να είχαμε θέσει επομένω το, πρόβλημα του ρόλου τη ε, Κεντρική Τράπεζα και τη παρέμβασή τη στην πρωτογενή αγορά. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκό, ένα ευρωπαϊκό ταμείο που ε, ε, εκδίδει ευρωμόλογα που μπορεί να ξαναγοράσει η Κεντρική Τράπεζα. Και μια και οι Βρετανοί δεν συμμετέχουν. Θα μπορούσαμε να είχαμε θέσει το θέμα τη εναρμόνιση τη δημοσιονομική, το πρόβλημα του κοινοτικού προπολογισμού και να προχωρήσουμε πραγματικά προ μια ομοσπονδιακή Ευρώπη που πολλοί από εμά θέλουμε. Ε, αυτό σημαίνει, συνθήκη, ε, σημαίνει συζήτηση για τη συνθήκη, σημαίνει τουλάχιστον συνέλευση. Και εγώ καταλαβαίνω αυτούς από ε, τους συντρόφους που λένε ότι όταν εκλεγούν πρόεδροι δημοκρατίας θα ξαναδιαπραγματευτούν τη συνθήκη. Ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Ήδη στην Αύκο το απόγευμα είχα συνταγματικές αντιρρήσεις για αυτή τη συμφωνία. Δεν έχει καθεστώς επίσημη συνθήκης. Είναι ιδιωτική συμφωνία μεταξύ μερικών και όχι όλων των χωρών. Και δεν σκοπεύω να επαναλάβω αυτά που είπα ξανά. Εκτός από το εξής, δεν θα ήταν σωστό, ίσως και παράνομο, να χρησιμοποιεί είτε η ψευτοκοινοτική αυτή μέθοδος για αυτόν τον σκοπό. Η ενιαία ισοτιμία για όλες τις χώρες δεν βολεύει όλες από αυτές. Και το ίδιο ισχύει και για τα επιτόκια, για 17 διαφορετικές οικονομίες. Καμιά φορά όμως ακούμε ότι αν κινηθούμε προς την Δημοσιονομική Ένωση ή την Πολιτική Ένωση, τότε κατά κάποιον τρόπο θα εξαφανιστούν αυτά τα προβλήματα και οι οικονομικές επικρίσεις δεν θα ισχύουν πια. Αλλά το γεγονός ότι πρόκειται για διαφορετικές οικονομίες που βρίσκονται παρόλα αυτά σε μια ενιαία οργάνωση δημοσιονομική είναι το πρόβλημα. Ακόμα και σε ένα κράτος μπορεί να υπάρχουν περιφέρειες με περισσότερα και άλλες με λιγότερα οικονομικά προβλήματα, ανεργία κλπ. Αυτό ίσχυε και το 30 παγκοσμίως στο Ηνωμένο Βασίλειο δεκαετία του 80 και ξανά του 90. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, ένα, ότι τα ενιαία κράτη έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν τις πιο καθυστερημένες τους περιοχές. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο αντιρρήσεις. Μία είναι ότι οι κυβερνήσεις πάντοτε έχουν την τάση να κάνουν, να το παρακάνουν σε αυτή την κατεύθυνση και ακόμη και αν κάνουν κάτι η δράση τους δεν λύνει πάντα το πρόβλημα. Η απάντηση δεν είναι νέα συνθήκη, αλλά οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, της Ευρωζώνης, να αλλάξουν το νόμισμά τους, να αλλάξουν την ισοτιμία και για, να μπορέσουν έτσι να έχουν εξαγωγές και να φύγουν, να βγουν από την κρίση. Δεν χρειάζονται οικονομικοπολιτικό ζουρλομανδία που θα τις οδηγήσει στην ανέχεια. Η υπερβάνς. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδροι, μάλλον. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια και η Ευρωπαϊκή ε, Κομισιόν δεν είναι πλέον ο θεματοφύλακας της συνθήκης, εμείς έχουμε την ευθύνη για το πώς διαχειριστούμε την προσεχή περίοδο. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι υπάρχει ένα συλλογικός πολιτικός κίνδυνος που όλοι, ή ρίσκο μάλλον, που όλοι αναλαμβάνουμε. Μπήκαμε σε μια συμβολική μάχη, δίνουμε μια συμβολική μάχη, αλλά κανένας δεν είπε ότι αυτό που υπάρχει σε αυτό το σχέδιο διαθεσμικής ή μάλλον διακυβερνητικής καλύτερα συμφωνίας δεν θα μπορούσε να γίνει εκτός των συνθήκων. Δίνουμε μια συμβολική μάχη λοιπόν. Δίνουμε μια συμβολική μάχη που διαιρεί τους Ευρωπαίους που μας οδηγεί σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας για να κερδίσουμε τι, κάτι το συμβολικό πάλι. Που πάει αντίθετα, εντελώς αντίθετα σε αυτό που χρειαζόμαστε. Γιατί κανένας δεν αμφισβητεί ότι χρειαζόμαστε λίγη δημοσιονομική πειθαρχία. Αλλά εδώ και πάνω από 10 χρόνια η Ευρώπη βρίσκεται κάτω από το δυναμικό ανάπτυξής της. Εδώ και δέκα χρόνια βρίσκεται κάτω από αυτό το δυναμικό. Γιατί, γιατί ε, επέβαλε αυτόν το μόνο, ε, ως μόνο κανόνα στις οικονομικές πολιτικές της το σύμφωνο σταθερότητας που θεωρώ ότι είναι μια παιδική φάση της, της ε, οικονομικής πολιτικής που είναι ανίκανο να λύσει τα προβλήματα ενός μεγάλου χώρου όπως η Ευρωζώνη. σε αυτή τη μάχη θα πρέπει να πάρουμε θέση. Καταρχάς, σε θεσμικό επίπεδο και απέναντι στις οικονομικές πολιτικές που θέλουμε να προωθήσουμε. Είναι δύο διαφορετικά μέτωπα, αλλά εδώ, σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο επίπεδα. Τώρα, για τη θέση του Κοινοβουλίου. Εγώ δεν έχω πολλές αμφιβολίες. Υπάρχει μια διαίρεση για το six-pack. Αν θυμάμαι καλά, ψηφίσαμε μια έκθεση και είχαμε και μία ειδική επιτροπή για την κρίση, όπου η συλλογική απάντηση που δώσαμε είναι, ήταν ότι για να βγούμε από αυτή την κρίση χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη κοινοτική μέθοδο. Και όχι λιγότερη Ευρώπη, λιγότερη κοινοτική μέθοδο όπως προβλέπει αυτή η συμφωνία που μας προτείνουν. Υπάρχει ένα πραγματάκι που με εκπλήσει ε, σε όλα αυτά που λέγονται. Και στην έκθεση για την κρίση, αλλά και στην έκθεση για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, είπαμε δύο φορά. Δύο φορέ ότι αν κάνουμε μια νέα μεταρρύθμιση των συνθήκη, δεν θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια μια συνέλευση. μας παγίδευσαν. Ε, και μας λένε ότι πρόκειται όχι για πραγματική συνθήκη της Ένωσης αλλά για συμφωνία, υποτίθεται. Εγώ δεν νομίζω ότι η σημερινή συνθήκη μας επιτρέπει να λύσουμε όλα τα προβλήματα της ζώνης ευρώ. Αλλά τότε το πραγματικό ερώτημα είναι το ε, ερώτημα της ανοιχτής συνέλευσης. Για να, μπουν όλα στο τραπέζι. Είναι αυτό που μας λέει ε, ο, ο Γκίφερ Χόφστατ. Θα κάνουμε κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο. Το μικρό είναι αυτή η συμβολική μάχη που πάει ενάντια στα όσα χρειαζόμαστε. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Τώρα για τα νομικά, μια κουβέντα ακόμα. Οι εκπρόσωποι μας βρίσκονται σε δύσκολη θέση, το ξέρω. Ε, θα πρέπει να λειτουργήσουν στα πλαίσια μια εντολή που έλαβαν από τη διάσκεψη των Προέδρων. Εγώ να σα ρωτήσω το εξή. Θα σα δώσουμε πολλού οδικού χάρτε. Αλλά δεν μπορείτε να δεχτείτε ένα κείμενο. Δεν μπορούμε να παίξουμε τον, των διασωτών αυτής της προσπάθειας και να δεχτούμε την αναφορά στο σύμφωνο Europlus ε, που είναι 20 φορές χειρότερο το σύμφωνο σταθερότητας. Είναι ένα χαρτί που το γράψαν στην Τοβίλ μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας που το έχει ανακυκλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν συζητήθηκε ποτέ δημοκρατικά σε κανένα κοινοβούλιο. Σας λέω ειλικρινά. Εντάξει, κατάλαβα τι είπατε τρεις φορέ και στι τρει παρεμβάσει σας. Μιλάτε, εστιάστε περισσότερο στα θεσμικά θέματα. Αλλά μην αγνοείτε το περιεχόμενο. Τι υπάρχει από πίσω από όλα αυτά τα χαρτιά. Γιατί αυτό που υπάρχει από πίσω είναι η επιδίνωση των δεινών που γνωρίζει η Ευρωζώνη από την αρχή της. Ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν διαφορές στην ε, ε, ανταγωνιστικότητα, ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες και δυναμικό ανάπτυξης κάτω από αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ότι δεν αντιμετωπίζουμε το, τη δημοκρατική, δημογραφική συγγνώμη, πρόκληση και την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά την εντολή που σας δόθηκε, για αυτή τη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, να δούμε πώς θα πορευτείτε. Γιατί η συμβολική μάχη που μας προτείνεται είναι ότι δεν σας άρεσε το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά το ενισχύουμε το six-pack και θα το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Και ο κανόνας θα γίνει τώρα 0,5% δημοσιο έλλειμμα. Με έναν τρόπο που κανένας δεν ορίζει πώς. Ευχαριστώ. Για τερμάκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαίρω αυτούς τους τρεις σοφούς που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο. Δεν είναι εύκολη η δουλειά τους, αλλά ελπίζω να πετύχουν. Τρία σχόλια. Πρώτον, τονίζω την κοινοτική μέθοδο. Δεύτερον, Νομίζω ότι όσο σημαντική και να είναι η δημοσιονομική πειθαρχία και η οικονομική διακυβέρνηση, υπάρχει και το θέμα του πώς πρέπει να προετοιμάζονται τέτοιου είδους δηλώσεις όπως την πούμε. Διότι τώρα θα ήθελα να σας πω πως ένας λόγος της κρίσης είναι και ότι όλες οι διασκέψεις και κορυφής έχουν προετοιμαστεί πολύ άσκημα. Κανείς δεν έχει πια εμπιστοσύνη και δεν ξέρει ακριβώς τι έχει αποφασιστεί. Γιατί και τρεις μέρες μετά τη συνάντηση ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι είπανε. Τα άρθρα λοιπόν που αφορούν τι πρέπει να κάνουμε πριν και μετά τη συνεδριάσεις είναι πολύ σημαντικά. Έπειτα. Τρίτο σχόλιο. Θα ήθελα να δειχτούμε όλοι, να φανούμε όλοι ρεαλιστές, δηλαδή για την δημοσιονομική πειθαρχία νομίζω ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι ρεαλιστικά, δηλαδή το 0,5 το μισό της διαρθρωτικού ελλείμματος δεν είναι ρεαλιστικό. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μετά από μερικά χρόνια. Πάλι τα κράτη-μέλη θα ξεπεράσουν ό,τι και να έχει γραφτεί. Αν δούμε τους αριθμούς τώρα, μόνο τρεις χώρες μέλη εκπληρούν πληρούν τα κριτήρια. Άρα, στο εξής, πρέπει να έχουμε άλλα κριτήρια που να μπορούν να τα τηρήσουν όλες ή σχεδόν όλες οι χώρες. Τώρα δεν μπορούν. Και αν χρειαστεί τα επόμενα δύο-τρία χρόνια να αρχίσουμε να επιβάλλουμε και πρόστιμα, δεν είναι σωστή μέθοδος αυτή. Ευχαριστώ. Θυμάμαι ότι και για την εξάμετρο χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο πριν περάσουμε στην ουσία. Με ξεπερνούσαμε τα μεσάνυχτα κλπ. Ελπίζω να μην γίνει και εδώ έτσι. Επόμενη από την εικόνη Μαρίαν Τάισεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους τρεις εισηγητές. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ε, πήγε σε μια περιπέτεια την οποία καλό είναι να συνεργαζόμαστε ε, αν η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή. Είναι πάρα πολύ σοβαρή όμως γιατί βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που ρίει αυτή τη στιγμή ε, το ευρώ αναταράσσεται στα θεμέλια του και το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας τίθεται, γιατί πολλά έχουν αλλάξει και πολλά πρέπει να αλλάξουν. Οι αρχαίοι κρατών κυβερνήσεων όμως αποφάσισαν ότι θέλουν μια νέα συνθήκη. Τι να κάνουμε. Να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Τώρα, να μείνουμε εκτός νηφώνος δεν έχει νόημα, δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Πρέπει να συνεργαστούμε και πρέπει να συνεργαστούμε εφιώς. Και αυτό που έχουμε επιτάπητος τώρα που το διάβασα με τα νομικά μου μάτια, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ένα συνοθήλευμα, αν μπορώ να το πω αυτό. Εάν στο πανεπιστήμιο ένας από τους φοιτητές μου μου έδινε ένα τέτοιο έγγραφο, οπωσδήποτε θα τον έκοβα. Είναι πραγματικά ένα συνοθήλευμα εμένα που βρήκαν από εδώ, βρήκαν εκεί και τα συνένωσαν. Και όταν ρωτήσει κανένας αυτό είναι ένα κείμενο με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε, είναι πραγματικά ένα κείμενο που θα μας δώσει τη λύση. Ελπίζω, τι να πω, ελπίζω ότι θα υπάρξει λύση. Πρέπει όμως να εργαστούμε με το κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή και η συμβουλή μου προς τους τρεις εκπροσώπους μας είναι ότι θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο ό,τι μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρο. Γιατί αυτό ήταν ένα, μια συμβολική κίνηση ό,τι μπορεί να επιληθεί μέσα στη συνθήκη που υπάρχει να λυθεί εκεί. Ό,τι μπορεί εκτός εκεί. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πολύ σύντομα. Και ο κύριος ε, Φερνόσπατ είπε ότι αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στη συνθήκη. Ναι, θα πρέπει πραγματικά να μπει μέσα στη συνθήκη όσον αφορά και την ιδέα και τη μέθοδο. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορεί να προσαρμοστεί. Εμείς δηλαδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε την κοινοτική μέθοδο, έχουμε τα θεσμικά όργανα, τρία-τέσσερα πολιτικά θεσμικά όργανα. Λοιπόν, ό,τι υπάρξει σε αυτή τη νέα συνθήκη θα πρέπει να εξεταστεί βάσει αυτών, προτού ενταχθεί στη συνθήκη. Ένας από τους τρεις εκπροσώπους μας αναφέρθηκε στην ρήτρα του ηλιοβασιλέματος, στη Sunset Clause. Εντάξει, αλλά θα πρέπει αυτόματα να είναι ε, σε σχέση με αυτά που πρόκειται να γίνουν στη συνθήκη. Γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν ακόμα. Και κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε ρεαλισμό. Το ανέφεραν οι προλήσαντες και εγώ θα το ζητούσα. Και σας παρακαλώ μην προσπαθείτε να πείτε στους πολίτες ότι με ένα τέτοιο μικρό κείμενο, μια συνθηκούλα αν μπορώ να την πω έτσι, θα λυθεί η κρίση. Όχι. Η κρίση είναι πολύ πιο ευρεία, όχι μόνο δημοσιονομική πειθαρχία και πολλά άλλα. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε ρεαλιστές και να είμαστε ρεαλιστές έναντι των πολιτών στην παρουσίαση που θα τους κάνουμε. Και θα ήταν καλό στρατηγικά νομίζω να ζητήσουμε να βρούμε εταίρους μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί λέμε πάντα για το ντουέτο Γερμανία-Γαλλία, οι οποίοι υποτίθεται ότι προωθούν ε, το χορό. Αν χορέψουν προς το κατεύθυνση καλά είναι, δεν λέω. Αλλά είναι καλό να αναζητήσουμε και άλλους εταίρους, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν συμφωνούν. Έτσι νιώθω τουλάχιστον, δεν μπορώ να το αποδείξω. Έχω την εντύπωση ότι οι άλλες χώρες δεν μπορούν να πούνε τίποτα σε αυτές τις συνεδριάσεις, παρόλο που θα ήταν καλό να τις ακούσουμε, ίσως θα μπορούσαμε να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο. Να αναζητήσουμε δηλαδή εταίρους και συμμάχους στις μικρές και στις μεγάλες χώρες μέλη, να τους κάνουμε προτάσεις που δεν μπορούν να κάνουν εκείνοι και έτσι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την εργασία εδώ, τον τρόπο εργασία στο Κοινοβούλιο, έχουν από τα εξής. Έχουμε του τρει σοφού, να του πούμε έτσι. Είναι τρεις άντρες, καλοί όμως, καλοί. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά πώς θα συνεχίσουμε εδώ την εργασία μας. Πώς θα εκφράσουμε δηλαδή τις απόψεις μας. Ακούσατε τι είχαμε να πούμε, δεν είναι πάντα ξεκάθαρα τα μηνύματα αυτά που ακούτε. Ποια θα είναι η εντολή που θα έχετε στη συνεδρίασή σας και πώς θα γίνει και η συνεννόηση μαζί μας και προς τους δύο συμπρόεδρους έχω να πω ότι νομίζω για την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου προβλέπεται μια συνεδρίαση, δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, θα ήθελα να μου το πείτε. Κουρμάι. Well Μπράβο σας. Ήταν σημαντικό που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση σήμερα. Το βασικό ορόσημο είναι το νομοθετικό πακέτο, το περίφημο six-pack και η εφαρμογή του. Και είμαι ικανοποιημένη που η βασική δουλειά έγινε επί Ουγγρικής Προεδρίας. Πιστεύω ότι οι κανόνες του six-pack είναι επίκαιροι, ε, μπήκαν σε ισχύ λίγες μέρες μετά την τελευταία Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Οι πέντε κανονισμοί και η μία οδηγία που φτιάχνουν το πακέτο των έξι είναι το μεγαλύτερο πακέτο για την εφαρμογή της ε, οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ένωση, από τη δημιουργία του ευρώ. Μας δίνει μια άμεση λύση, ε, μια δέσμη εργαλείων, ούτως ώστε να υπάρχει ε, πειθαρχία για να παρεμποδιστεί μια νέα κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω ορισμένου και λυπάμαι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλησε μια διακυβερνητική συνθήκη λόγω του ότι δεν συμφώνησαν και 27. Αντί να μπορέσει να δεχτεί την πρόταση που, μια πρόταση που ήταν πολύ πιο προσεκτική. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοινοβουλίου, ε, αναγνωριζόταν και ενισχυόταν εκεί. Το αποτέλεσμα όμως είναι, είναι μια διακυβερνητική συνεννόηση που βασίζεται πολύ που θα έπρεπε να βασίσετε περισσότερο στην κοινοτική μέθοδο. Τα μέτρα θα πρέπει να αποφασίσετε μέσω δευτερογενής ε, νομοθεσίας, αλλά μόνο με τη συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, παρακολούθησα την κάλυψη του τύπου ε, των τελευταίων ημερών και πιστεύω ότι οι οικοτολογίες σε ορισμένα μέσα, ότι η συνθήκη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αυτό είναι λάθος. Αντίθετα από αυτά που λένε ορισμένα ΜΜΕ, το αποτέλεσμα τη ε, συνόδου είναι καλύτερο από ό,τι φαίνεται ε, προ ό,τι όψεω. Υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποι μα θα υλοποιήσουν του στόχου του. Και του έχουμε καλή τύχη γιατί έχουν μεγάλε προκλήσει μπροστά του, όπω και όλοι μα. Μια ισχυρή Ευρώπη. Είναι μια Ευρώπη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε για ανάπτυξη και θέσει απασχόληση. Ε, γι' αυτό υποστήριζω την ιδέα του κ. Ντόντο. Χρειαζόμαστε σταθερότητα αλλά χρειαζόμαστε και ανάπτυξη. Ευχαριστώ, καλά Χριστούγεννα και ελπίζω ε, να μην σας κοιμήσει το six pack. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ich meine... Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ κατά βάση δεν θα ήθελα να πω πια τίποτα, γιατί η ανησυχία μου ε, αυξάνεται λεπτό με λεπτό. Έχουμε ένα θέμα. Ε, η διάσκεψη πήρε μια απόφαση. Η αγορά δεν αγόρασε πάνω σε αυτή. Δεν αγόρασε. Δεν, δεν αντέδρασε η αγορά. Ούτε οι πολίτες αντέδρασαν γιατί υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο αυτό που αποφασίστηκε μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια και να οδηγήσει σε βελτίωση κατάστασης. Και εμείς συζητάμε τώρα την απάντηση. Έχει κανένα την εντύπωση ότι αυτή θα είναι η απάντηση που θα α, εξαλείψει την ε, δυσπιστία και την έλλειψη της εμπιστοσύνης στις πολιτικές αποφάσεις. Όχι, όχι. Όποιο επιχείρημα και αν χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, εμείς βρισκόμαστε ακόμα πριν την απόφαση της διάσκεψης κορυφής και όχι στην στιγμή της εφαρμογής της απόφασης. Δεύτερος σημείο. Η Περβός Περές είπε ότι πρόκειται για μια συμβολική μάχη. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή συμβολικές μάχες. Σε αυτή τη στιγμή την οποία αναφέρθηκε και η Μαριάν Τάισεν. Δεν χρειαζόμαστε συμβολικές μάχες, ούτε επιτρέπεται να παίξουμε το παιχνίδι αυτό με τις συμβολικές μάχες. Ούτε εμείς θα πρέπει να συμβάλλουμε σε ε, συμβολικές μάχες. Χρειαζόμαστε σοβαρά και αποφασιστικότητα. Τρίτον, θα το πω ξεκάθαρα. Υπάρχουν κάποιε αιτίε για την κρίση. Τρει. Το ευρώ στηρίζεται σε ένα πόδι μόνο και ε, φοβηθήκαμε να πάρουμε την πολιτική ευθύνη για το ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτή την πρόταση θα αναλυφθεί η πολιτική ευθύνη για το ευρώ. Ναι. Επίσης, δεν λάβαμε υπόψη σοβαρά τους δικούς μας κανόνες γιατί δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους εαυτούς μας. Και γι' αυτό δεν τηρούμε και τους κανόνες. Αυτή η πρόταση θα οδηγήσει σε συνεπή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και υιοθετημένων οδηγιών, ναι ή όχι. Ναι. Και μπο... είμαστε ευάλωτοι από εκβιασμούς της αγοράς, των κερδοσκόπων και από εμά τους ίδιου ως πολιτικοί. Εγώ δεν θα αναφερθώ ε, στο ότι μας τραβάνε από τη μύτη η Γαλλογερμανία εδώ πέρα. Και όταν λέει ο κύριος ε, Φερχόφστατ ότι πρόκειται για ένα διακανονισμό βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, μακροπρόθεσμη λύση δεν επιτρέπεται να είναι. Θέλω γιατί για τη μακροπρόθεσμη λύση χρειαζόμαστε συνέλευση. Αλλά ούτε και βροχή πρόθεσμη μπορεί να είναι γιατί η στερή αυτών υπαρχόντων. Το six-pack και το κοινοτικό δίκαιο πάνε πολύ πιο μακριά. Τελευταίο σημείο λοιπόν. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι θεματοφύλακας των συνθήκων και που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας διαπραγματευόμαστε πάνω σε μια πρόταση του Συμβουλίου και όχι βάσει μιας πρότασης του ιδίου του Κοινοβουλίου, ούτε μια πρόταση της Κομισιόν. Απαιτώ κατεπηγόντως πρόταση που θα απορρέει από την... αυτό που είπε ο Παρόζο, εγώ είμαι η οικονομική κυβέρνηση. Πού είναι η πρόταση της Κομισιόν βάσει αυτού του ρητού εμείς είμαστε η οικονομική κυβέρνηση. Και πού είναι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του ρητού εμείς είμαστε η δημοκρατική νομιμότητα και χωρίς εμάς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Διαπραγματευόμαστε μια πρόταση με την οποία δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη μέθοδο των τροπολογιών και έτσι βρισκόμαστε σε αμυντική στάση. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε επί ίσης όρης ξέρω τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Τέσσερα σημεία έχω ακόμα να παρουσιάσω. Για μένα είναι σίγουρο ότι η συνθήκη αυτή θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει αντίφαση όσον αφορά το περιεχόμενο θα πρέπει να συμπληρώνει και να εμβαθύνει και να βελτιώνει τις συνθήκες της Λισαβόνας και να εξαλείφει τις αδυναμίες της. Δεύτερον, δεν επιτρέπεται να αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την συναπόφαση. Θα πρέπει να διευρύνει τις δυνατότητες συναπόφασης. Και τρίτον, η Κομισιόν θα πρέπει να παραμείνει θεματοφύλακα της συνθήκες, έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και το Συμβούλιο δεν είναι κυβέρνηση, είναι νομοθέτης. Τέταρτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επίσης νομοθέτης. Το Συμβούλιο είναι απέναντί μας, όχι τα εθνικά κοινοβούλια. Και οτιδήποτε λοιπόν επανεθνικοποιεί την συνθήκη δεν είναι σύμφωνο με τις αρχές του σώματος. Θα πρέπει με αυτές τις προτάσεις να δούμε ότι με τα στοιχεία που έχουμε δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Σούλτς. Ευχαριστώ. Πολλά ελέγχθησαν. Θα μπορούσα να συμφωνήσω σχεδόν 100% με τον προλαλήσαντα, πράγμα που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εδώ στο σώμα. Τέλο πάντων, θα ήθελα να αναφέρω και τρει άλλε πηγέ. Η δική μου ομάδα, σύμφωνα, δεν είναι ομόφωνη. Αλλά θα ήθελα να σα πω ξεκάθαρα, ναι, στην κοινοτική μέθοδο, σαν απαραίτητο στοιχείο της συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε λύση. Η οποιαδήποτε λύση δεν θα υπάρξει όμως θα πρέπει να ξανεξετάσουμε κανένα πόσο όπως είπε ο μακροπρόθεσμα όχι βάσει της ισχύω αυτή, της, προτάσεις, της πρότασης που έχει υποβληθεί και ο χαρακτηρισμός αυτού του συνοθηλεύματος του νομικού έγινε ήδη. Μακροπρόθεσμα όμως θα μπορούσαμε να περάσουμε στη σκέψη προς τα που θέλουμε να κινηθούμε. Και εδώ βρισκόμαστε στην πραγματικότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σήμερα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να κοιτεχτούμε στον, κατέ, στον καθρέφτη και να ρωτηθούμε προτιθέμεθα τα σφάλματα που υπάρχουν στις συνθήκες μέχρι στιγμής που επιτρέπουν χάσμα μεταξύ της νομιματικής ένωσης και της οικονομικής ένωσης των κοινωνικών πτυχών και των ε, πτυχών της απασχόλησης προτιθέμεθα λέω να αναπτύξουμε την ένωση αυτή. Δηλαδή εκτός από τη σταθερότητα το ρόλο της ε, Κεντρικής Τράπεζας και του ΣΥΚΣΠΕΚ χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι που θα πρέπει να μας κάνει να ακολουθήσουμε την πραγματική ευρωπαϊκή κοινωτική πολιτική. Περισσότερη Ευρώπη λοιπόν θα απάντηση προς την κρίση. Δεύτερον, έχουμε και μια πολιτική κρίση. Έχει δίκιο ο Άντριου Νταφ που το είπε. Βρισκόμαστε στην πιο βαθιά και σοβαρή κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν την ε, ξεπεράσουμε με αυτές τις ε, ε, ε, διακοσμητικές αν θέλετε διορθώσεις. Όχι. Μονάχα εάν ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών, των πολιτών, της κοινή γενικά. Και αν δεν κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, και αυτό είναι νομίζω και τμήμα της εντολής της ε, διαπραγματευτικής ομάδας, και αν δεν πούμε ξεκάθαρα ότι εμείς επιμένουμε στην κοινωτική μέθοδο, επιμένουμε σε μια κοινοτική βάση και δεν επιτρέπουμε εκτός από τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει και διακυβερνητική νέα συνθήκη με εθνικές συμφωνίες γιατί αυτό πραγματικά θα οδηγήσει στην καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μακροπρόθεσμα δεν θα οδηγήσει ούτε σε βελτίωση οικονομική, ούτε κοινωνική, ούτε περιβαλλοντολογική, ούτε τίποτα. Και τρίτο σημείο θα πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη στιγμή το ποιο είναι ο στόχο τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θέλουμε δηλαδή μόνο να διασώσουμε το ευρώ ή μήπω θέλουμε και μια κοινωνική Ευρώπη, μια περιβαλλοντολογική Ευρώπη και μια ειρηνική Ευρώπη. Γιατί φοβούμε ότι αν δεν καταφέρουμε να απαντήσουμε ξεκάθαρα στην κρίση αυτή προωθώντας την ε, κοινοτική μέθοδο, θα ξαναπεράσουμε σε εθνικοποιήσεις που θα καταστρέψουν μια ένωση 60 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους κινδύνους που θα ενέχεται κάτι τέτοιο. Και αν δούμε πως η τέταρτη ισχύ της κοινωνίας οδηγεί σε ε, διαμάχες μεταξύ των εθνών, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε προς την άγουσα που διακυβεύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό οι τέσσερις προτινόμενες ε, ε, μέθοδοι για την ομάδα διαπραγμάτευσης που υπέβαλε ο συνάδελφος Κάρας είναι νομίζω η σωστή βάση. Ευχαριστώ. E- Κυρία Σάντσες Περσέντο, η τελευταία μιλήτρια από την ΕΚΟΝ. Ο κύριος μάλλον. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Είμαστε στο μέσο μιας κρίσης οι κεντρικέ τράπεζε των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόσουν την, ε, τη συμφωνία. Θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τα μέτρα. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, να υπάρξει οικονομικό συντονισμός, η συνθήκη μας το επιτρέπει απόλυτα. Έχουμε την δευτερεύουσα νομοθεσία για να το πράξουμε. Μία συνθήκη θα μπορούσε να έχει νόημα Καταρχάς, αν θέλουμε να δεσμευτούμε πραγματικά σε ψηλό επίπεδο και να πούμε ότι θα σημειώσουμε πρόοδο με μεταβίβαση κυριαρχίας τότε μία συνθήκη μπορεί να είναι χρήσιμη. ιδίως αν τα κρατημέλη δεν μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία της αναθεώρησης. Μία συνθήκη μπορεί να έχει νόημα, αλλά σε αυτή τη συγκυρία είναι χρήσιμη μία συνθήκη. Αυτό είναι το ερώτημα. Η συνθήκη θα λέει ότι θα πάμε σε μία δημοσιονομική και οικονομική ένωση. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, όχι διακοσμητικές προσπάθειες. Όχι. Επιμένουμε στο six-pack. Πρέπει να μιλήσουμε για οικονομική διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για ακυρώσεις. Θέλουμε ένα ευέλικτο σύστημα, ώστε αυτή η μεταφορά κυριαρχίας να γίνεται χωρίς να περνάμε κάθε φορά από την ομοφωνία. Είναι μια ευκαιρία που έχουμε. και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια κοινοτόμα μέθοδο. Δηλαδή, η Κομισιόν θα μπορούσε να εμπλακεί στη διαδικασία και τελικά να έχουμε μια συνθήκη πλάς. Θα πρέπει να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μας χρειάζεται. Ο κύριος Σταβαρέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Γκουλάχ, η Σιλβί Γκουλάχ, μα είπε ότι θα δημιουργήσουμε ένα τέρας. Φυσικά δεν είναι τεχνικό όρο όρος, όρος τέρας. Ο, ο τεχνικός όρος που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το double ganger. Αυτό το πλάσμα που εμφανίζεται, που έχει κρίση προσωπικότητας και που διχάζεται. Έχουμε το, τον κλασικό άνθρωπο με την ε, σύνθετη προσωπικότητά του και έχουμε και αυτό το πράγμα το οποίο έχει μονομανίες. Έχουμε ήδη την Ένωση και με την ε, συνθήκη θα είχαμε την ε, Doppelganger που λένε οι Γερμανοί. Ένα πλάσμα που είναι τρελαμένο με τους δημοσιονομικούς κανόνες για την διατήρηση του ευρώ. Σε αυτό το το μυθιστόρημα Dr. Jekyll και κύριο Hyde όμω, θα υπάρχουν πάντα θύματα. Και το πρώτο θύμα θα ήταν το κοινοβούλιο το οποίο θα αποκλειόταν από την όλη διαδικασία. Έχω λοιπόν να κάνω μία ερώτηση στους τρεις συναδέλφους στα πλαίσια αυτής της παρέμβασής μου. Ποια στιγμή Από ποια στιγμή και μετά λέμε στα κράτη-μέλη, στην Κομισιόν, που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και από ό,τι φαίνεται δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν υπερασπίζεται τις συνθήκες. Από ποια στιγμή θα πούμε θα κάνουμε μια, θα δημιουργήσουμε μια συνέλευση ούτω ώστε να κρατήσουμε την ένεση και να μην υπάρχει αυτός ο διχασμός της προσωπικότητας. Πώ θα αποφύγουμε η Ένωση να σκοτώσει την Ένωση. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το, το, μόρφωμα, αυτό το πλάσμα με τη διχασμένη προσωπικότητα που θα σκοτώσει ουσιαστικά τον εαυτό της. Είχατε πει ότι είχαμε πει να είμαστε σύντομοι, ναι, αλλά και εγώ τους άκουσα όλους και Έχω ένα πολύ σύντομο πράγμα από μία έκκληση. Εγώ είμαι από μικρή χώρα εκτός Ευρωζώνης και θέλω να μπει σε αυτήν. Η διέρεση όμως στο εσωτερικό της Ευρώπης είναι καταστροφική. Γι' αυτό παρακαλώ κύριοι, ακόμη κι αν τελικά δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε, προσπαθήστε να διευκολύνετε τα πράγματα για αυτούς που θέλουν να μπουν στην Ευρωζώνη και μη βάζετε περαιτέρω φοηραγμούς και εκδικητικά αισθήματα γιατί χρειαζόμαστε ενωμένη πραγματικά Ευρώπη και εδώ έχουμε μία πολύ πραγματική αποστολή να εκτελέσουμε. Πολύ ωραία. Οι τρεις παρατηρητές μας θα συνοψίσουν τώρα. Συνοψίσουν. Σω θα πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά με την οποία θα παρέμβω, ο κύριο Φερχόφστατ πρώτο, ας πούμε. Πώ μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο τώρα, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε. Ας πω καταρχήν, ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η συμφωνία δεν θα λύσει την κρίση. Δεν θα ρυθμίσει τα τη κρίση η απόφαση του Ντράγκη σήμερα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ξεκινήσει μια πιστοτική γραμμή 200 ε, εκατομμύρων ευρώ με 1%, ε, με 1 επιτόκιο θα πετύχει περισσότερα από αυτό, από αυτό το κείμενο. Μπορούμε να υπερβούμε την κρίση με τουρισμό, με χρήματα και με hardware. Μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με αυτή τη συμφωνία. Αλλά η συμφωνία θα υπάρχει σε λίγες εβδομάδες. Χωνέψτε το. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά που είπατε θα κάνουν να εξαφανιστεί αυτό το κείμενο. Όχι, θα υπάρχει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξή. Μπορούμε να πούμε δεν μας ενδιαφέρει, δεν μπαίνουμε θέση, δεν μπαίνουμε μέσα στην ιστορία ή προσπαθούμε να το, βελτιώσουμε. Εγώ νομίζω πρέπει να κάνουμε το δεύτερο, να το βελτιώσουμε. Για να αποφύγουμε αυτό το, το τέρας ή τη διχασμένη προσωπικότητα που είπατε. Ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να πάμε στο δικαστήριο. Μπορούμε να σταματήσουμε να νομοθετούμε, επειδή δεν συμφωνούμε με αυτό το κείμενο. Α πούμε στο Βέλγιο τα συνδικάτα αυτό κάνουν, τα στυλώνουν. Τρίτον, μπορούμε να πάρουμε δική μας πρωτοβουλία για να αλλάξουμε τη συνθήκη με δική μας πρωτοβουλία. Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτοί κάνουν αυτό, εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε διάφορες δυνατότητες, έχουμε διάφορα εργαλεία που μπορούμε να επιλέξουμε. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε στις διαπραγματεύσεις και να πούμε μπορούμε να κάνουμε κάτι κατά αυτού του κειμένου να σταματήσουμε να νομοθετούμε, να κάνουμε μια δική μα πρωτοβουλία για αλλαγή τη συνθήκη, α τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα χαρτιά για να βελτιώσουμε το κείμενο από την... Το βελτιώσουμε. Ίσως είναι μια ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουν, να βάλουμε πράγματα που δεν θέλουν. Φερρυπίν, η ιδέα της ε, συνθήκη, τη ρήτρα Sunset. Ότι όλα μπορούν να μπουν, δηλαδή, τελικά να ενσωματωθούν στη σημερινή συνθήκη. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δεύτερον, δεύτερη ιδέα. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητε. Δεύτερη. Έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο εφετήθηκε σήμερα νομίζω, έτσι. Για τα, σύμφω... για τα ομόλογα σταθερότητα. Έχουμε το κείμενο της Κομισιόν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νομική βάση. Μπορούμε. Έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία. Η σημερινή συνθήκη δεν επιτρέπει κάτι, άρα να δημιουργήσουμε μια άλλη νομική βάση. Άλλο παράδειγμα, άλλη δυνατότητα. Όλοι μπορούν να είναι κατά, αλλά αν δεν καταλαβαίνετε ότι, ότι πρέπει να έχουμε κοινά ομόλογα όταν έχουμε κοινό νόμισμα, τότε είστε τυφλοί. Οι, οι Αμερικάνοι το κάνανε το 18ο αιώνα. Το 1790 ο Χάμιλτον το έκανε. Ξυπνήστε. Ήτανε Χάμιλτον εναντίον Τζέφερσον. Κέρδισε ο Χάμιλτον. Το κάνανε οι Αμερικάνοι το 18ο αιώνα. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε, άντε, 200 χρόνια μετά στην Ευρώπη. Μια άλλη ιδέα. Μιλούσαμε για το σύμφωνο Europlus και όλα τα σχετικά. Ή θα τα βγάλουμε όλα αυτά από τη συμφωνία. Το Σέγγεν δεν έχει καμία σχέση. Είναι η λύση δεμήνυμα, minima, Να τα βάλουμε όλα εκτός η άλλη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε το κείμενο για να πετύχουμε διάφορα πράγματα, να ενισχύσουμε τη συνεργασία. Γιατί με αυτή τη συμφωνία, αν ε, επιβάλλουμε την ενισχυμένη συνεργασία, τότε μπαίνει και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Έτσι βάζουμε ξανά μέσα στο σύστημα τους δύο αυτούς παίχτες, με την ενισχυμένη συνεργασία. Γιατί αυτό προβλέπεται στη συνθήκη. Μπορούμε να πάμε και πιο μακριά. Γιατί να μην είστε φιλόδοξοι σε αυτά που προτείνουμε τις επόμενες εβδομάδες στο τραπέζι. Θέλετε οικονομική διακυβέρνηση ή μάλλον όχι θέλετε ενισχυμένη συνεργασία. Φτιάξτε μια συμφωνία να χρησιμοποιήσουμε το 333 της συνθήκης και να πάμε από την ομοφωνία στην ενισχυμένη πλειοψηφία αμέσως για αυτά τα θέματα. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ο Πορτογάλος συνάδελφος είπε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό θετικά για να πετύχουμε πράγματα που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να πετύχουμε. Θέλουν συνθήκη. Εμείς θέλουμε κάποια πράγματα. Ας τα βάλουμε στο τραπέζι. Τέλος. Τελευταίο παράδειγμα. Για το 273. Χρησιμοποίησαν το 273. Ε, πότε δεν έχει να χρησιμοποιηθεί, ναι. Είναι θέμα χωρών. Ε, χρησιμοποιείται όταν μια χώρα είναι αντίον μιας άλλης στο δικαστήριο. Ας βάλουμε και την Κομισιόν. Μπορούμε να το κάνουμε. Ας βάλουμε εκεί μέσα και την Κομισιόν. Θέλουν ενισχυμένη πλειοψηφία. Θέλουν την αντίστροφη ενισχυμένη πλειοψηφία. Ας χρησιμοποιήσουμε την διαπραγμάτευση, ούτω ώστε να βάλουμε μέσα την πραγματική οικονομική διακυβέρνηση. Αλλά όλα αυτά υπό τον όρο ότι θα πέσουν, θα μπουν στην ε, σημερινή συνθήκη τελικά. Αλλιώ θα έχουμε το τη διχασμένη προσωπικότητα τελικά. Επίσης, να σας πω ότι ο Έλμαρ είναι πολύ καλός. Ροκανίζει έτσι τις θέσεις των κρατών μελών. Βλέπει που ε, ανταποκρίνονται θετικά έτσι και πάει λίγο παραπέρα. Είναι πολύ έξυπνος. Και είναι, είναι πολύ ευγενικό απέναντι σε αυτέ τι χώρε που λένε θέλουμε το Α, το Β. Προσπαθεί να δημιουργήσει συμμαχίε με διάφορε χώρε. Ακούσαμε διάφορε χώρε στι παρεμβάσει του που λέγανε τα ίδια ακριβώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ίδια με αυτέ. Μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιε συμμαχίε λοιπόν. Πότε θα ξαναβρεθούμε Τώρα, να διοργανώσουμε μια τέτοια ξανά μια συνεδρίαση, σύντομα. Ούτω ώστε να έρθουμε εδώ πέρα και να τα ξαναπούμε μαζί σας, να έχουμε μια επαφή. Thank you. Ευχαριστώ. Θα τα πω Ιταλικά αυτή τη φορά. Γιατί... Και αργά. Ας μιλήσει Ιταλικά λοιπόν. Πρώτο θέμα το οποίο τέθηκε. Η συνευθύνη, συνυπευθυνότητα. Να τα πω ξεκάθαρα. Εμείς ήμασταν επικριτικοί και για τη φύση αυτού του επιλεγέντος εργαλείου και μάλιστα με εξέπληξε το γεγονός ότι πολλές αντιπροσωπείες είπαν το ίδιο με μένα. Καμία δεν είπα, ή μάλλον σχεδόν καμία δεν είπε ότι αυτή η επιλογή είναι οι καλύτεροι. Σχεδόν οι περισσότεροι είπαν ότι καλύτερα θα ήταν να είχαμε κάνει κάτι άλλο, ε, να είχαμε βρει κάτι άλλο. Αυτό έχουμε τώρα μπροστά μας. Ε, επικρίναμε ακόμα και το περιεχόμενο όμω του εγγράφου. Όπως είπε ο Γκί, το καθήκον μας είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και για να μειώσουμε τη ζημιά και για να καταστήσουμε αυτή την ε, συνθήκη, η συμφωνία αν θέλετε, ευκαιρία αν θέλετε για την μελλοντική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως και πιθανότητα μιας ήτας, ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι για μένα ισχύει αυτό που είπαν πολλοί άλλοι, ότι επιφυλάσσονται να αξιολογήσουν την, την όλη ιστορία, το όλο αποτέλεσμα στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Το είπαν πολλοί αυτό αυτό θα πρέπει να ισχύει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν είμαι συνυπεύθυνο λοιπόν. Δεν αισθάνομαι συνυπεύθυνο. Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και μετά θα αξιολογήσουμε, όχι εμεί, οι τρει, το Κοινοβούλιο το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νομική φύση του κειμένου μας. Θετικό. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το γεγονός ότι το άρθρο 2 του σχεδίου της συνθήκης κρατάει την αρχή της ισχύω της κοινοτική νομοθεσίας, του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου. Λέει ότι καμία ε, διάταξη αυτής της συνθήκης δεν ισχύει σε περίπτωση που έρχεται σε αντίφαση με πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν το διαφυλάσσουμε. Καλό είναι και πρέπει να να κρατηθεί αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Ότι το κείμενο αυτό δεν συνάδει με αυτή τη διατύπωση, με αυτή τη διάταξη. Η εξήγηση που μας δόθηκε για τη διαφορετική φύση των διαφόρων διατάξεων από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου ήταν ότι υπάρχουν δύο ειδών διατάξεις, λέει. Πρώτη, πρώτος τύπος, πρώτη μορφή διάταξη. Μια πολιτική δέσμευση να συμπεριφερθούμε με συγκεκριμένο τρόπο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οκ, okay. Ε, θεμητό. Τα κράτη μπορούν να αποφασίσουν να λειτουργήσουμε συγκεκριμένο τρόπο απέναντι στα θεσμικά μας όργανα. Δεύτερον, η ε, υιοθέτηση ψηλότερων προτύπων σε σχέση με αυτό που προβλέπει η συνθήκη στα πλαίσια της δευτερογενούς νομοθεσίας. Τώρα εδώ μπαίνουμε σε θολά νερά, σε λεπτές ισορροπίες, σε λεπτά πράγματα. Ε, γιατί ουσιαστικά γίνεται και μια ποιοτική αλλίωση αυτών των ε, στάνταρ αυτών των προϋποθέσεων. Πέρα από την ποσοτική αλλαγή, από το που φτάνουμε δηλαδή στο 0,5 του ελλείμματος, αλλά αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για εθνική επαλήθευση της, α, ε, του σεβασμού των διατάξεων. Έχουμε δηλαδή κάποια μέτρα πιο ε, αυστηρά και κάποια μέτρα πολύ πιο ελαστικά. Αυτή η υποχρέωση διόρθωσης για μας είναι βασικό θέμα. Και αυτό μπορεί να γίνει με, με διάφορους τρόπους. Εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ότι οι, πρώτες, οι του πρώτου είδους θα πρέπει να υπερισχύσουν και να υπάρχει αυτή η πολιτική δέσμευση μέσω της κοινωτικής νομοθεσίας να ε, σεβόμαστε διάφορες αρχές και δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και αλληλεγγύη και ανάπτυξη και δημοκρατία. Που πρέπει να είναι όχι αφηρημένες έννοιες, αλλά στοιχεία χωρίς τα οποία δεν μπορεί να βγει η Ευρώπη από την κρίση. Επίσης, πώς η Κομισιόν μπορεί να παίξει το ρόλο του υποκινητή, αν θέλετε. Πώς μπορεί να κάνει προτάσεις. Προτάσεις ε, κανονισμού, προτάσεις ενισχυμένης συνεργασία. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ή το έκανε πολύ κατακαιρματισμένα με τις δύο προτάσεις κανονισμού με βάση το, 100, το άρθρο 136. Ελπίζουμε αυτή η διαδικασία, η διαπραγματευτική, να αναγκάσει την Κομισιόν να, γίνει, να δραστηριοποιηθεί λιγάκι, να κουνηθεί λιγάκι. Ε, στον πρώτο γύρο, με δυσαρέσκεια άκουσα που πολλά πέρα από το Κοινοβούλιο, είναι πολύ πιο αποφασιστικά στο να υποστηρίξουν το ρόλο της Κομισιόν από ότι η ίδια η Κομισιόν. Ήταν εντελώς αδρανής η Κομισιόν στην πρώτη ας πούμε φάση, στον πρώτο γύρο. Εν συνεχεία βέβαια όταν προέκυψε διαφωνία ότι δεν υπήρξε δηλαδή, παθητική ας πούμε, υπερψήφιση αυτού του α, σχεδίου κειμένου, αλλά αποφασίστηκε να γίνει σοβαρή συζήτηση, τότε εντάξει, άν και η Κομισιόν και έγινε πιο δραστήρια. Ελπίζουμε τώρα αυτό να μεταφραστεί και σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίε της Κομισιόν. Φυσικά και εμείς ω Κοινοβούλιο μπορούμε να πάρουμε τέτοιε πρωτοβουλίε. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε μια συνέλευση. Αλλά τώρα είμαστε εδώ γιατί δεν υπήρχε ομοφωνία. Ούτε καν για την ε, αναθεώρηση του πρωτοκόλου 12. Δεν νομίζω τουλάχιστον λοιπόν ε, με αυτό το δεδομένο ότι βραχυπρόθεσμα θα ήταν μια βιώσιμη διαφυγή από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ε, ότι όλες αυτές οι διατάξεις μπαίνουν στην ε, συνθήκη, όπως ακριβώς είπαν οι συνάδελφοι. Και με την επιφύλαξη των προνομίων και των υποχρεώσεων που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα πρωτοβουλία, μπορεί να κάνει προτάσει, θέλει να, το ασχίσει. Εξάλλου το Σεπτέμβριο είχα προτείνει σε μία έκθεση πρωτοβουλία ακριβώ το ίδιο. Ίσως καλό θα ήταν να το είχαν δεχτεί, να είχαν δεχτεί τότε αυτή την έκθεση οι πολιτικές ομάδες, ούτως ώστε να ξέρουμε ξεκάθαρα τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο και τι δεν μπορεί να κάνει για τις συνθήκες. Επίσης, ε, αυτά που λέγονται για πολιτικό ρεαλισμό, για προσπάθεια να οικοδομήσουμε συμμαχίε, όλα αυτά είναι, ισχύουν απόλυτα. Και ελπίζουμε να μπορούμε να βασιστούμε στου ε, συναδέλφου για να δημιουργήσουμε συμμαχίε με τι εθνικέ αντιπροσωπείε. Τέλο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό όλα αυτά σημαντικά που άκουσα να μεταφραστούν και σε γραπτέ προτάσει βέβαια. Το συντομότερο και γενικέ προτάσει, αλλά και πολύ συγκεκριμένες μετροπολογίε. Γιατί τώρα είμαστε σε φάση, α, στη φάση τη κατάρθων εξέταση. Πρέπει να κάνουμε τη γενική συζήτηση για τη φύση της, τη φύση της συμφωνίας, αλλά εν συνεχεία θα μπούμε σε μια πολύ λεπτομερή εξέταση, άρθρο προς άρθρο. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει κάπως να επιταχύνουμε κι εμείς. Πρέπει να εντοπίσουμε πολύ συγκεκριμένα τι τροπολογίες θέλουμε, ε, και πώς θα οικοδομήσουμε συμμαχίε για να περάσουμε αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο κύριο Μπρόκ. Κλείνοντα αυτή τη συζήτηση. Πρόεδρε. Πολλά ευκταία. Μπορεί να το υπογραμμίσει κανένα, αλλά θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Πρώτον, τα κράτη-μέλα είναι η μόνη κυρίαρχη οποιασδήποτε συνθήκε. Μπορούμε να αναλάβουμε όποιε πρωτοβουλίε θέλουμε, αλλά δεν αναλέγει τίποτα. Είτε για την τροποποίηση τη διοίκηση τη Αβώνα πρόκειται, είτε για διακυβερνητική συμφωνία. Η μόνη κύριε τη συνθήκη είναι τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό οι πρωτοβουλίε που μπορούμε να κάνουμε σε θεσμικό επίπεδο είναι περιορισμένε. Δεύτερον, τι θα κάνει το πρωτογενέ δίκαιο πρέπει να δώσει ένα νομικό πλαίσιο, να δώσει νομικής βάσης, αλλά δεν μπορεί οι πολιτικές μάχες να περάσουν στο πρωτογενές δίκαιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε άλλα επίπεδα. Δευτερογενές δίκαιο, Φερρυπίνη. Και γι' αυτό συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα ελέγχθησαν, ότι αυτή η πρόταση της ηθίκης δεν λύνει τα ε, οικονομικά προβλήματα. Αυτό δεν το λένε καν και εκείνοι που θέλουν αυτή τη συνθήκη. Γιατί χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα. Παραδείγματο χάρη ε, κάποιου ε, κανονισμού στι ε, χρηματαγορέ. Και γι' αυτό χαίρομαι ότι η βρετανική πρόταση ομοφωνία για τις ε, δημοσιονομικές αγορές, αλλαγές μάλλον, θα πρέπει να δίνεται μόνο με ομοφωνία δεν πέρασε γιατί αυτό θα κατέσει αυτή την εσωτερική αγορά. Και το δεύτερο πρόβλημα, ο διακανονισμό των οικονομικών αγορών θα ήταν το μόνο σημείο στο οποίο θα είχαμε συγκεντρώσει την προσοχή μας. Δεν ήταν δυνατόν 27 χώρες να ε, θελήσουν την αλληλική συνθήκη. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα πολλές αντιπροσωπείες είπαν ότι αυτή η βάση διακυβερνητικής σύμβασης είναι μονάχα η δεύτερη σε ποιότητα λύση. Και έτσι θα πρέπει να την εμπλούσουμε κιόλας. Και να μην ε, ζητήσουμε πολλά από αυτή. Υπάρχουν δύο σημεία για τα οποία χρειαζόμασταν, θα χρειαζόμασταν αλλαγή της συνθήκης. Ή τρία μάλλον. Το ένα είναι ο χρυσός κανόνας το δεύτερο είναι αντίστροφη πλειοψηφία. Παρόλο που και εκεί υπάρχει κάποια διαφωνία κατά πόσο χρειάζεται πράγματι. Και το τρίτο είναι ενδεχομένω μια νομική βάση για τα ευρωομόλογα. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα διακανονίσουμε με τη σημερινή συνθήκη τη αγώνα. Όλα τα υπόλοιπα. Μια από αυτή η διακυβερνητική βάση είναι πάντα προβληματική για το Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσουμε καταρχήν να μην είναι πολύ επιτυχής αυτή η διαδικασία. Γιατί άμα προσεχώς 27 δεν μπορούμε να ε, πετύχουμε ομοφωνία για μια αλλαγή της συνθήκης, αλλά 9 κράτη θα αρκούν για να, πετύχουμε, να πετύχουν μάλλον μια τέτοια συνθήκη εκτός, τότε θα έχουμε χάσει από σκοπιά κοινοβουλίου. Γι' αυτό πρέπει να αποδώσουμε σημασία η νομική βάση που υπάρχει είναι μία αυτοϋποχρέωση των κρατομελών. Τίποτα άλλο. Και εκεί θα πρέπει να αρκεστούμε και θα πρέπει να φροντίζουμε αυτή η αυτοϋποχρέωση να μην περάσει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν θα μπορεί να ε, έχει τα ε, να προηγηθεί της ε, συνθήκης, να μην άπτεται των δικαιωμάτων στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα μπορούμε να καταδείξουμε την αξιοπιστία μιας τέτοιας απόφασης πράγμα που προσπαθήσαμε με μία μικρή ε, επιτυχία σήμερα το πρωί, κάποια στιγμή να το θέσουμε αυτό στην ε, κοινωνική νομοθεσία ή να το εντάξουμε συνθήκη στην πρώτη ευκαιρία ή με μια ρήτρα ήλιο βασιλόμητος ή κάτι παρόμοιο. Κατόπιν. Αυτή είναι η βάση που παρουσίασε η Μαριάννα αυτη ειναι η βαση που παρουσιασε η μαρια ταισεν και όταν κάρας βέβαια. Κατόπιν, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η κοινωτική μέθοδος είναι η μέθοδος της δυνατότητας δράσης διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμότητας. Γιατί η διακυβερνητική αλλιώς σημαίνει ομοφωνία και καμία ε, και καμία συμμετοχή δημοκρατική. Ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο ακρόαση όμω, όχι στην απόφαση. Αυτό πρέπει να πούμε στου αδέλφου στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Εμεί οι τρει και άλλοι βέβαια. Θα πρέπει να πάμε στις σύμμαχες κυβερνήσεις και να δημιουργήσουμε συνασπισμούς για να προστατεύσουμε τη θέση μας. Και κάτι άλλο. Ίσως μία συνεδρία λιγότερη στις Βρυξέλλες και ο καθένας από εμάς να πάει στο εθνικό του κόμμα, στο εθνικό του βουλή, στην εθνική κυβέρνηση και να πει «Για ακούστε, μην έχουμε δεκάρικες εδώ στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Βασοβία, στο Βερολίνο». Αλλά εργασία. και να υπάρχει ανησυχία ότι μπορούν όλα να πάνε στραβά για να επιτευχθεί έτσι βούληση συμβιβασμού για τη θέση αυτή. Αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερο σημείο. Πρωτοβουλίες. Ακούσαμε. Μα άμα έχουμε μία σειρά θέματα που ε, μπορούν να λυθούν στη δευτερογενέ δίκαιο, γιατί δεν αρπάζουμε την Κομισιόν εδώ για να τα λύσει τα θέματα αυτά. Να πούμε, θέλετε να δυναμώσετε το σύμφωνο σταθερότητα με την αντίστροφη πλειοψηφία. Για ελάτε το Κομισιόν, για πέστε μα κάτι για τον επόμενο γύρο για το σύμφωνο σταθερότητα, ε, Μπορούμε να βάλουμε το ευρώ μόνο, δεν το έχουμε εκεί κάποια άλλα. Η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκουνηθεί Σήμερα είπανε θα σας υποστηρίξουμε. Με πολύ πυγμή, μετά που είχε τελειώσει η συνεδρίαση όμως. Όπως όταν λέμε, όταν χρειαστεί να κουβαλήσουμε τον κυνηγό στο κυνήγι, το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ θετικό. Λοιπόν, Κάτι παρόμοιο θα πρέπει να κάνουμε την Κομισιόν, να τη δοκουνήσουμε. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα πρέπει να βγάζουμε για αυτούς το φίδι από την τρύπα. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Λοιπόν, σαφείς ορισμοί, ο στόχος, κοινοτική πολιτική, σύμμαχοι και συνασπισμοί με τους συναδέλφους στις Εθνικές Βουλέ και στα κόμματα και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του στο δικό τομέα. Εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιες μάχες ε, καθυστερημένες για το six-pack. Αυτό το κάνουμε στον επόμενο γύρο της νομοθεσίας. Όχι αυτά που δεν υπάρχουν στο six-pack, δηλαδή να μπουν συνθήκη. Γιατί σας προειδοποιώ, αυτά δεν θα είναι πια υπό επίδραση και έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να σου πούμε, αυτά θα πρέπει να διακανονιστούν στο six-pack. Την επόμενη φορά θα πρέπει να είναι καλύτερο το six-pack αυτό. Βέβαια, διαφορετικά ε, κόμματα έχουν διαφορετικές απόψεις και οι απόψεις αυτές θα παραμείνουν. Θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαμάχη, ναι, μεταξύ μας, καθημερινά. Όχι να τα μεταφέρουμε αυτά σε άλλο επίπεδο, γιατί το επίπεδο στο οποίο θα τα μεταφέρουμε δεν είναι το δικό μας επίπεδο. Ναι, ίσως έχεις δίκιο. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Αλλά αυτή η συνθήκη δεν είναι ο τόπος που θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Γιατί μόνο με εξοικονομήσεις δεν πλούσε ποτέ κανένα τα χρέη του. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, να εξεταστεί το θέμα της ανάπτυξης κλπ. Με ισορροπία. Αλλά ε, ε, σκεφτόμαστε πώς θα βάλουμε τον όρο ανάπτυξη εκεί μέσα. Ο Ρομπέρτο το κοιτάνε, αλλά θα πρέπει να δούμε και μέχρι πού θα πάμε για να μην το κάνουν διακυβερνητικό θέμα τους. Θα ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τι διατυπώμουν, πού το διατυπώμουν για να μην στραφεί εναντίον μας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε μια τέτοια υποέλεγχο στρατηγική. Εκτός από ε, το πρωτοβουλίες που θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε ο καθένας στην πατρίδα μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες ε, που είναι σημαντικές για μας ε, αύριο. Δεύτερον, αν έχει κανένας μια πρόταση πώς θα πρέπει να αλλάξει κάποιο άρθρο. Μια πρόταση, μια λέξη, όχι μακρά κείμενα, αλλά αν έχετε κάποια ιδέα να μας το υποβάλλετε γραπτό σας παρακαλώ. Και όταν έχουμε μια τέτοια συνεδρίαση ξανά, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ θα πάω στην ομάδα μου και οι συναδελφοί θα κάνουν το ίδιο. Θα παρουσιάσω τα πράγματα, ίσως πρόεδρε, πρόεδρε, Αυτέ οι δύο επιτροπέ που θα μπορούσαν να ορίσουν ίσω μια, μια μικρή ομάδα, συγγνώμη, 8-10 ατόμων, που με ένα τηλεφωνηματάκι μπορούμε να του συνενώσουμε, να συνεδριάσουμε και να δώσουμε τι πληροφορίε που υπάρχουν από τη συνεδρίαση. Όχι όλοι ίσω αυτή η ομάδα, αλλά ε, μια μικρή ομάδα εργασία που θα μπορούμε να σε εγκαλέσουμε σε δύο ώρε, για να έχουμε έτσι αυτή την ε, επιστροφή των ιδεών που όχι μόνο θέλουμε να σας δώσουμε, αλλά τη χρειαζόμαστε εμείς για να έχουμε την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ξανάρθετε βέβαια και θα οργανώσουμε και εμείς συνεννοήσεις. Στο άρθρο 7 θέλω να σχολιάσω κάτι, όπου γίνεται λόγος για την αντίστροφη πλειοψηφία στην εξάμετρο του Six λέγαμε, αναφέραμε το άρθρο 283β, όχι 238α. Άμα, δηλαδή 72% αντί για 65. Ήθελα να το αποσαφηνίσω να το ξέρετε. Γιατί χρειάζεται εδώ συνέπεια. Σας ευχαριστώ όλους και λυπούμε λοιπόν που τόσο πολύ. un di lavoro και εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεδρίαση αυτή. Στην ΑΦΚΟ έχουμε έκτακτη συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου. Θα έχουμε πολύ δουλειά τότε, αλλά ίσως να βρούμε κάποιο χρόνο. Βρούμε κάποιο χρόνο μου λέει η γραμματεία ότι μπορούμε ίσως να εισακούσουμε αυτά που είπατε εσείς. Ε, Ευχαριστούμε, χαίρετε. Davvero. Buon Natale da parte di questa Presidenza. <laughs> Buon Natale. Soprattutto...